Good morning, dear colleagues. Let's start. Ε, καλημέρα σας. Ε, να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Και θα μιλήσω λιθανικά. Λοιπόν, η μερίσια διάταξη, της οποίας το πρώτο θέμα είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εντάξει, εγκρίνεται. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Οπότε συνεχίζουμε. Δεύτερο, ανακοινώσεις ε, της Προέδρου, μόνο μία. Να σας ενημερώσω για τις αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Το σημείο 9 της ημερήσία διάταξης θα προταχθεί της ψηφοφορίας. Και το περνάμε τώρα στο σημείο 3 της μέρης διάταξης. Έχουμε εδώ λοιπόν μια έκθεση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στα εξωτερικά, στις εξωτερικές σχέσεις συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα γίνει συζήτηση για το θέμα αυτό, απλώς μια ενημέρωση. για το χρονοδιάγραμμα εξέτασης αυτής της έκθεσης. Και μάλιστα δεν είναι έκθεση, είναι γνωμοδότηση, η οποία θα υποβληθεί 23 Φεβρουαρίου την επόμενη εβδομάδα και η προθεσμία είναι στις 29 Μαρτίου μέχρι τις 6 ε, ώρα το απόγευμα και θα υποβληθεί στις 23 Μαρτίου και θα ψηφίσουμε 8 και 9 Απριλίου στη δική μας Επιτροπή ενώ η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ θα γίνει 23-24 Μαΐου και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Αυτό λοιπόν είναι το χρονοδιάγραμμα εξέτασης ε, της ε, γνωμοδότησης αυτής ε, και να περάσουμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Προϋπολογισμός για το 2017 εντολή για τον τριμερή διάλογο. Ο εισηγητής είναι ο Γιέντς Γκάια από πλευράς της Επιτροπής Προϋπολογισμών και μας ε, έχει επισκεφθεί εδώ. Ξέρω ότι θα επισκεφθεί όλες τις επιτροπές, ε, θα προσπαθήσει να ενημερωθεί για τις προτεραιότητες όλων των επιτροπών για να τις λάβει υπόψη στη διαμόρφωση της γενικής του θέσης. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή, ευχαριστώ κύριε Γκάι για την παρουσία σας. Ελπίζω να έχουμε μια καλή ανταλλαγή απόψεων. Να δώσω λοιπόν το λόγο στο Γιέννης Γκάια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα ξεκινώ το γύρο επισκέψεων ε, στις ε, κοινοβουλευτικές μας επιτροπές με την επίσκεψη στη δική σας επιτροπή κάποιος σας έψαχνε λέει κάποια κυρία μα εδώ είμαι λέει ο κύριος Γκάιερ τι έλεγα λοιπόν αρχίζω τις επισκέψεις επιτροπών με τη δική σας εδώ στην Επιτροπή Γυναικών θα πρέπει να συνεργαστούμε γιατί ο συνάδελφος ή ε, συνάδελφος ε, Νόιχελ ε, συμμετέχει στην ψηφοφορία. Θα είναι ενδιαφέρουσες οι διαπραγματεύσεις που επίκυνται για τον προπολογισμό του 2017 γιατί στην παρούσα συγκυρία η Ένωση αντιμετωπίζει μεγάλες δυσχέρειες. Όπως λέμε, ο προϋπολογισμός είναι πολιτική αποτυπωμένη σε στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τα νομοθετήματα που έχουμε και τη στήριξη των πολιτικών μας πρωτοβουλειών με κονδύλια. Παντού στην Ευρώπη ε, αντιμετωπίζουμε και συζητάμε την κρίση των προσφύγων η οποία όλο και περισσότερο οξύνεται και θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα απαιτηθούν πολλά κονδύλια, τα οποία όμως δεν έχουμε. Ε, στην κατηγορία 3 για την εσωτερική πολιτική έχουμε δαπανίσει 5 δις για να απαλύνουμε την κρίση του προσφυγικού και τα αίτια της και να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της. Την κατάσταση τη γνωρίζετε όλοι από τις ειδήσει. Οξύνεται συνεχώς η κρίση. Δεν μειώνεται. Βεβαίως μια μικρή ελπίδα είναι η κατάπαυση του πυρός στη Συρία, αλλά πέραν τούτου δεν. Άρα δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλλουμε ότι τα κονδύλια του προπολογισμού για το θέμα αυτό θα είναι περισσότερα, αλλά τα άρα τα υπόλοιπα λιγότερα. Και είχαμε χθε ε, μια πρώτη διαπραγμάτευση, την λεγόμενη ΕΑΡΙΝΗ διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και είναι κυρίως copy-paste. Πολύ λίγες αλλαγές δηλαδή ε, προτίθεται το Συμβούλιο να κάνει, έχει ήδη κάνει πολύ λίγες αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές για τον προπολογισμό του 2016 και μένουν σε αυτά που χρόνια τώρα λένε τα δύο θέματα που μας ε, βρίσκουν αντίθετους είναι κυρίως ότι οι πολιετής δημοσιονομικές ε, προοπτικές ε, αντιμετωπίζονται ως οι δέκα εντολές δεν μπορούν να φυγούν και δεν μας επαρκούν τα όρια που προβλέπουν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές εάν θέλουμε να έχουμε ουσιώδεις αλλαγές στον προπολογισμό. Το δεύτερο βασικό επιχείρημα του Συμβουλίου είναι ότι εντός ε, των ε, ανωτά των ωραίων που προβλέπουν οι πολιτείς προοπτικές θέλουμε να έχουμε και κάποια περιθώρια για να αντιμετωπίσουμε απρόβλεπτες καταστάσεις. Τι άλλο απρόβλεπτο μπορεί να προκύψει η Πολλά βέβαια. Τώρα αν είχαμε ε, τώρα την τα φύλλα δάφνης της πυθίας μπορεί και να ξέραμε. Αλλά για το 16 έχουμε πλήρως ούτως ή άλλως εξαντλήσει αυτά τα όρια. Χθες εγκρίναμε ήδη τον πρώτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 16, όχι επίσημα εντελώς, αλλά υπάρχει συμφωνία και αυτή η πρώτη αλλαγή του προϋπολογισμού του 16 πρώτα απ' όλα προβλέπει 100 εκατομμύρια βοήθεια άμεση για να βελτιωθεί η κατάσταση ε, στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Φύρων και για να ε, προσλάβει η Europol περισσότερο προσωπικό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο προϋπολογισμός του 16 έχει εξαντληθεί πλήρως ενώ αρχίζει το, ο τρίτος μήνας του 16 και χρειαζόμαστε ήδη συμπληρωματικό προπολογισμό. Δεν αλλάζουν λοιπόν οι προκλήσεις, αλλά το Συμβούλιο φέρεται σαν να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, σαν να είναι συνηθισμένη η κατάσταση και θέλει να παραμείνουμε στα προβλεπόμενα από τις δημοσιονομικές προοπτικές ανώτατα όρια. Γιατί τα αναφέρω αυτά. Γιατί η δική σας Επιτροπή ασχολείται με προγράμματα της κατηγορίας 3, εσωτερική πολιτική του προϋπολογισμού. Για το Δάφνη ισχύει αυτό, για άλλα προγράμματα που σας απασχολούν, για το φορέα, για την ισότητα των φύλων. Και βεβαίως ε, συμφωνώ απόλυτα με τις πολιτικές σας προτεραιότητες, τις κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Συμπεριλαμβάνεται ότι Επιθυμώ να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, αλλά θέλω επίσης να καταστήσω σαφές ότι οι δυνατότητες που θα έχουμε για τον προπολογισμό του 17 είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Γι' αυτόν το θέμα δεν είναι μόνο να εκφράσουμε όλοι τις επιθυμίες μας, αλλά να καταλάβουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα όλες οι επιθυμίες που θα προκύψουν από τις 20 επιτροπές του σώματός μας δεν θα μπορέσουν να γίνουν σεβαστές. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε προτεραιότητες. Αλλά γενικά ο προπολογισμό διαμορφώνεται έτσι που θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Το Συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ότι πρέπει να καθοριστούν προτεραιότητες. Βεβαίως, να καθοριστούν. Ο Ολλανδός ε, υπουργό, όταν το ρώτησα ε, τι εννοείται ακριβώς να θέσουμε προτεραιότητες, ισχύουν ή όχι πλέον οι στόχοι της Ευρώπης 2020. Δεν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Βεβαίως θέλουμε. Και στις οδηγίες που αποφασίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε ότι ιδιαίτερα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ε, φτώχεια των παιδιών. Φυσικά πρέπει να κάνουμε κάτι για να προκύψει περισσότερη απασχόληση και ανάπτυξη. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε κάτι ούτω ώστε το εύση να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως. Άρα θα πρέπει να θέσουμε ε, για εγγυήσεις αυτού του ταμείου μερικά δις ακόμη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στους καταβλισμούς προσφύγων, να καταπολεμήσουμε τα αίτια του προσφυγικού και κυρίως να ε, βοηθήσουμε τα πιο ευάλωτα τμήματα του προσφυγικού πληθυσμού, γυναίκες και παιδιά δηλαδή. Και πρέπει κάτι να κάνουμε για να, για να καταπολεμήσουμε αυτήν την θλιβερά υψηλή ανεργία των νέων. το Συμβούλιο ναι μεν εναντιμών αντιμετωπίζεται ενωμένο αλλά στην ουσία υπάρχουν βαθιές ε, ε, διαφορές. Είναι οι φίλοι της συνοχής, οι φίλοι της γεωργίας και οι φίλοι των επιστροφών. Και βεβαίως υπάρχει και διαφορά απόψεων για τον τρόπο χρηματοδότησης του ενωσιακού προϋπολογισμού. Άρα σε μεγάλο βαθμό όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα χειριστεί το προϋπολογισμό η Προεδρία. Όταν θα αναλάβει την Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο η Σλοβακία, που δεν είναι σαφές λόγω των εκλογών που μόλις έγιναν. Πολλά λοιπόν θα εξαρτηθούν από την επιδεξιότητα της Προεδρίας. Πώς θα καταφέρει να συνδυάσει τις αποκλίνουσες απόψεις στο Συμβούλιο και πώς, σε ποια βάση θα επιχειρήσει να συμφωνήσει μαζί μας. Δεν νομίζω ότι ο προπολογισμός θα είναι πολύ μικρότερος από τον Περισσινό. Και ε, ε, θυμάστε ότι ο περσινός προπολογισμό είχε φτάσει στα όρια των προοπτικών. Υπάρχει αυτός, ε, αυτό το περιθώριο για τα πρόβλεπτα, οπότε όσο περισσότερα πάρουμε φέτος για τον φετινό προϋπολογισμό για τα πρόβλεπτα, ε, όλα αυτά θα πρέπει να εξοικονομηθούν από τους επόμενους προϋπολογισμούς. Αν πάρουμε χρήματα από το αποθεματικό, τότε πρέπει να τα ξαναβάλουμε. Δηλαδή, αν ξοδέψουμε περισσότερα φέτο, θα πρέπει να ξοδέψουμε λιγότερα του χρόνου. Αυτό είναι το πλαίσιο που επιχείρησα να σα εξηγήσω και ε, με χαρά τώρα να ακούσω τα σχόλια και τι ερωτήσει σα. Σα ευχαριστώ όλοι, Και τώρα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και καταρχάς θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λαντσίλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση αυτή για τον προπολογισμό και για το γεγονός ότι μας ενημερώνεται και για τις προτεραιότητες. Είναι σημαντικό αυτό σε κάθε επιτροπή να τίθενται οι ανάλογες προτεραιότητες. Εμεί ε, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του 2017 έχουμε θέση από την Επιτροπή μας ε, πολλές προτεραιότητες. Καταρχάς, Μιλάμε για μια συνεκτική και σταθερή ε, διαμόρφωση των προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, γιατί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή το 2013 έθεσαν και προδιέγραψαν ότι σε όλα τα στοιχεία του προπολογισμού θα πρέπει να εντάσσεται και η διάσταση του φύλου. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια πολιτική ε, για την ισότητα των φύλων και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις φάσεις της κατάρτισης του προπολογισμού. Και οι διάφορες γραμμές του προπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ε, τη διάσταση του φύλου σε ό,τι αφορά τώρα τα διαστατικά ταμεία και τα επενδυτικά ταμεία. Σκοπός είναι η καλή κατάρτιση, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και για τις γυναίκες και για τα νεαρά κορίτσια. Τα μέσα λοιπόν αυτά θα πρέπει να προέλθουν από τις αντίστοιχε, από τα αντίστοιχα κεφάλαια του προϋπολογισμού, από τις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού, για να είναι ίσες οι ευκαιρίες που έχουν και οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια. για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά και τα θέματα μητρότητος ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν πρόκειται για μέτρα τα οποία αφορούν τις γυναίκες που ζουν στην Ήπεθρο. Οι γυναίκες, σε σχέση με τους άντρες, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ε, σε ό,τι αφορά τη φτώχεια. Αυτό λοιπόν έχει αναφερθεί ήδη. Για να καταπολεμηθεί λοιπόν η φτώχεια και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μητέρες με παιδιά, είναι σημαντικό να έχουν ευκαιρίες οι γυναίκες αυτές για την εξέβρεση εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω το να δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη γραμμή στον προπολογισμό της Ένωσης, στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προκειμένου να μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν τέτοιες πρωτοβουλίες όταν δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν ε, εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν δυνατότητε φύλαξη ε, των παιδιών και όταν ε, η απασχόληση είναι χαμηλή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προγραμματίσουμε και να σχεδιάσουμε λοιπόν τέτοια να τέτοια συστήματα για την υποστήριξη των γυναικών και ιδιαίτερα των περιστροπημένων γυναικών σε τέτοιε κοινότητε. Φυσικά το Κοινοβούλιο θέλει να καταπολεμήσει την ανεργία των νέων ιδιαίτερα Και σε ό,τι αφορά λοιπόν την πρωτοβουλία για την νεολαία, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν αρκετά κονδύλια. Να σεβαστούμε επίσης και την ισότητα σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου για τις γυναίκες και τις ε, κοπέλες. Ένα άλλο θέμα σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση του προγράμματος DAFNE. Αναφέρθηκε και αυτό. Και αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Από το 2013 μέχρι το 2020 το πρόγραμμα DAFNE δεν είναι ξεχωριστό πρόγραμμα, αλλά αποτελεί ένα συγκεκριμένο στόχο ενός ευρύτερου προγράμματος σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του πολίτη και την ισότητα. Ως εκ τούτου, τα κονδύλια ενδεχομένως να διακυμαίνονται σε ό,τι αφορά το ύψος του, γιατί υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς ναι, των κονδυλίων από τον ένα στόχο στον άλλο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει επαρκή κονδύλια το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει στεφτεί με ιδιαίτερη επιτυχία παρεπιπτόντως και θα πρέπει λοιπόν να λάβει πιο μεγάλη χρηματοδότηση. Για φέτος προβλέπονται ε, κάτι περισσότερο από 14 εκατομμύρια για το πρόγραμμα Daphne, το οποίο είναι λίγο παραπάνω από αυτά που προβλέπονταν για το 2014 και 2015. Όταν το πρόγραμμα Daphne είχε ξεχωριστεί η γραμμή οι δεσμεύσει για το πρόγραμμα ε, Daphne ήταν 18 εκατομμύρια για το 2011 και μάλιστα πάνω από 20 εκατομμύρια για το 2011. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει να προβάλλεται αυτό το όνομα Daphne σε όλες ε, τις διαστάσεις γιατί είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο το πρόγραμμα και μάλιστα τώρα με την ε, μεταναστευτική κρίση θεωρώ ότι το πρόγραμμα Daphne θα πρέπει να βοηθήσει τις γυναίκες και να λάβει και πιο πολλά κονδύλια. Κάτι άλλο τώρα πώς βοηθούμε τις ε, γυναίκες πρόσφυγες και τις ε, γυναίκες ετούντες άσυλο σε ό,τι αφορά την κατάσταση των προσφύγων, των γυναικών προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο ζήτησε πιο πολλά κονδύλια για να δοθεί καλύτερα η διάσταση του φύλου σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κρίση. Προτείνουμε να ε, προωθηθεί και το πρόγραμμα Οδυσσέας και το πρόγραμμα Δάφνη για να αντιμετωπίσουμε με καλύτερο τρόπο την τρέχουσα κατάσταση και να προστατεύσουμε τις γυναίκες πρόσφυγες. Τα κονδύλια που διατίθενται στις κοινωνικές οργανώσεις, στις οργανώσεις για την παρακολούθηση των δικαιωμάτων είναι και αυτά εξαιρετικά σημαντικά. ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, σε ό,τι αφορά την χρήση των ε, χρηματοοικονομικών μέσων, όπως ε, τα μέσα που αφιερώνονται στη μετανάστευση και στην ενσωμάτωση και εδώ θα πρέπει να επιμείνουμε. Ένα άλλο θέμα ενδιαφέρον είναι το Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων. Είχε ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο στα πλαίσια του Ιδρύματος αυτού για την ε, βία μεταξύ των φύλων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθούν επαρκή κονδύλια στο Ίδρυμα αυτό και να υπάρχει και αρκετό προσωπικό, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Αυτά αποτελούν τις προτεραιότητες μας για τον προπολογισμό του 2017 και φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι θα καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Πιστεύουμε δε ότι ακόμα και αν υπάρχουν προβλήματα στον προπολογισμό, αυτό που ζητάει η Επιτροπή μας, αυτά που ζητάει η Επιτροπή μα δεν μπορούν να αγνοηθούν και θα πρέπει να ενταχθούν στον προπολογισμό του 2017. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ eh, Jag har lyssnat noga på vad du σας ευχαριστώ πολύ. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα μας είπατε για τον προϋπολογισμό. Μην το πάρετε προσωπικά, αλλά εγώ ανησυχώ πάρα πολύ. Έχω την αίσθηση ότι από τη μια πλευρά μας λέτε ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις προσδοκίες μας και από την άλλη λέτε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ε, μπει σε όλες τις πολιτικές το gender mainstreaming και τα λοιπά. Μα, ε, ανησυχώ γιατί βλέπω τον τρόπο με τον οποίο η, η Κομισιόν ιεραρχεί τα κοινωνικά ζητήματα και πώς ε, αντιμετωπίζει τα θέματα ισότητας χωρίς να μας υποβάλει μια στρατηγική περί ισότητας των φύλων, το περιορίζει σε ένα έγγραφο εργασίας εσωτερικό Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα, έχουμε την αίσθηση ότι ο προπολογισμό μα είναι εξαιρετικά εκτεθειμένο λόγω των όσων συμβαίνουν και κυρίω λόγω τη προσφυγική κρίση. Τα θέματα τα κοινωνικά ξέρουμε ότι θα είναι φτωχό συγγενή. Όλοι γνωρίζουμε πω δεν είμαστε νομοθετική επιτροπή. Ξέρουμε ότι στη διάρκεια των ετών που είμαστε εδώ, εγώ είμαι εδώ, εδώ και 12 χρόνια και αγωνιζόμαστε για τα ζητήματα τη ισότητα κάθε φορά ώστε να μπουν στην ημερήσια διάταξη. Και το έχουμε καταφέρει σε κάποιο βαθμό, αλλά χρειαζόμαστε για να το στηρίξουμε. Γι' αυτό και ανησυχώ πάρα πολύ όταν βλέπω τις πιθανές εξελίξεις για την ισότητα των φύλων και την πιθανότητα να οπισθοχωρήσουμε εδώ πέρα, να οπισθοδρομήσουμε μάλλον. Τι θα γίνει με εκείνα τα ζητήματα που αφορούν τα γυναικεία δικαιώματα. Δεν πρόκειται μόνο για την ισότητα αυτή καθ' αυτή, αλλά και για δικαιώματα που, ε, που αφορούν το παιδί, γιατί συχνότερα είναι οι γυναίκες που ασχολούνται με τα παιδιά και εσείς ο ίδιος αναφέρετε το παράδειγμα της παιδικής φτώχειας. Έχουμε ένα σωρό στόχους λοιπόν. Έχουμε τους στόχους ε, του 2030 όπου η Δυτική Ευρώπη φέρει μέγα μέρος ευθύνης. Ξέρουμε όμως ε, ταυτόχρονα ότι το Συμβούλιο ακόμα και αν έχει αναφέρει τα θέματα της συνθήκης της Λισαβόνας και όλες τις στοιχές που ε, αναφέρονται εκεί και λένε τι ωραία και τι καλά αλλά στην ουσία χρήματα για να στηριχθούν όλα αυτά δεν δίνουν. Μήπως λοιπόν θα πρέπει διαφορετικά να χωρίσουμε το προπολογισμό. Μήπως πρέπει να εξετάσουμε το μίσο που δαπανώνται πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή και να ανακατανείμουμε πόρους από αυτά σε άλλα ζητήματα γιατί δεν νομίζω πως τα, κράματα, τα κάτι μέλη θα δώσουν χρήματα περισσότερα για τον προπολογισμό. Αυτά είναι και με αυτά πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Πάντως το θέμα είναι πως τα θέματα φύλου, τα θέματα ισότητας εν γέννη, τα θέματα που αφορούν τις μειονότητες είναι αυτά που θα υποφέρουν. Γιατί σε αυτό το σώμα πάντοτε η προτεραιότητα έχει αγορά. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόντι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ε, πολύ ωραία που σε βλέπουμε σήμερα εδώ. Χαίρομαι. Συνήθως σε βλέπω στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Απλά θέλω να αναφέρω κάποια σημεία που ήδη ε, έχουν αναφερθεί, ε, αλλά και να αναφέρω και κάτι νέο, δηλαδή όταν βλέπουμε τον προϋπολογισμό και τις επενδύσεις για δουλειές και για ανάπτυξη, συχνά παραμελούμε τις επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, που είναι ωστόσο κομμάτι της ανάπτυξης ε, της ατζέντα ε, για την ανάπτυξη και τις ε, θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει να δούμε και για τη φροντίδα των παιδιών, πράγμα το οποίο έχει αντίκτυπο στην παιδική φτώχεια. Είναι τομείς που θα πρέπει να μας απασχολήσουν και να τους τονίσουμε, να τους δώσουμε έμφαση. Κάτι άλλο που ήδη ανεφέρθη, αλλά που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι η στήριξη για το πρόγραμμα Δάφνη. Γιατί σε καιρούς λιτότητας τα κράτη-μέλη ξαφνικά η προστασία για τις γυναίκες και η βία κατά των γυναικών είναι κάτι που καλό θα ήταν να γινόταν, αλλά όχι κάτι που οφείλει, που πρέπει να γίνει. Ενώ αυτά τα προγράμματα είναι εξαιρετικά πολύτιμα και από οικονομικής άποψης μπορούν να σταθούν αυτά τα προγράμματα ακόμη. Κάτι ακόμα που νομίζω πρέπει να ενισχυθεί είναι όταν εξετάζουμε την κατάσταση των προσφύγων να πούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξεταστεί συγκεκριμένα η κατάσταση των γυναικών και παιδιών προσφύγων και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν προγράμματα στοχοθετημένα σε αυτούς, ώστε οι γυναίκες αυτές να μπορούν να στηριχθούν και να ενταχθούν στα προγράμματα. Ιδιαίτερα και όσον αφορά τις ε, κοινωνίες υποδοχής των προσφύγων. Ε, και κάτι ακόμα το οποίο είναι κοινό στις συζητήσεις για τον προπολογισμό, είναι η μέτρηση των ε, αποτελεσμάτων ε, performance budgeting, δηλαδή προπολογισμό με βάση τις επιδόσεις, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Και το κατά πόσο μέσα σε όλα αυτά ε, μπορεί να συμπεριληφθεί και προπολογισμό με βάση το φύλλο. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι αποδίδει ο προπολογισμό για το 51% του πληθυσμού και μετράται αυτή η απόδοση. Μετράτε ο προπολογισμό και για στις επιδόσεις του για τις γυναίκες. Ε, Ačiū, ponia Mūdė. Ε, ir dabar norėčiau pranešėjus suteikti žodį, pono Gėriui. Μάλιστα, και τώρα να δώσω το λόγο πάλι στον εισηγητή, στον κύριο Γκάιερ. Yeah, Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις παραβάση σας. να περιοριστώ σε τρία ζητήματα. Και εγώ δεν έχω παρατηθεί από τις ελπίδες μου να καταφέρουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν παραπάνω χρήματα στον προϋπολογισμό. Το πρόβλημα του ε, λοιπούς προϋπολογισμού αφορά όλες τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεν γίνεται συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο που να μην θέτω το θέμα αυτό. Και σίγουρα έχουμε καλά επιχειρήματα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Και εισαγωγικά μίλησα για μία τριχοτόμηση, αν θέλετε, του Συμβουλίου γιατί έτσι διαμορφώνονται η στάση των κρατών μελών σε ό,τι αφορά και την προθυμία τους και τον ανοιχτό χαρακτήρα που δείχνουν έναντι του προπολογισμού. Και οι κυβερνήσεις των δύο χωρών από τις οποίες προερχόμαστε δεν είναι από αυτές που θέλουν να δώσουν απαραίτητα πιο πολλά χρήματα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και έτσι λοιπόν δεν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε και πολλά πράγματα από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν δεν καταφέρουμε λοιπόν να έχουμε πιο πολλά χρήματα στον προϋπολογισμό, το θέμα είναι πώς μπορούμε να δαπανίσουμε με πιο σόφρονα τρόπο τα χρήματα αυτά που έχουμε. Δεν θέλω να υπονοήσω ότι πρέπει να ανησυχούμε και ότι το θέμα της ισότητας των φίλων θα παραμεριστεί και θα αγνοηθεί, γιατί υπάρχει μια σαφής πλειονότητα, πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υπέρ των θεμάτων αυτών και νομίζω ότι πάντα τα θέματα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Και σίγουρα θα ληφθούν όλα αυτά τα θέματα υπόψη στη συζήτηση στον προπολογισμό. Η Δάφνη, το πρόγραμμα Δάφνη. Στα προγράμματα κατηγορίας 3 σίγουρα θα έχει προτεραιότητα και πιστεύω ότι το όλο πρόγραμμα έχει αρκετά προηγουμένα κονδύλια περιορισμένα γιατί είναι τόσο σημαντική η πολιτική στόχη που περιλαμβάνει. Τόσο σημαντική είναι η στόχη αυτή που θα άξιζαν πραγματικά να λάβουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Και εδώ πραγματικά θα σας υποστηρίξω. Αλλά δεν θα χρησιμοποιούσα, όπως πρότεινε η συγγετρία, να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Daphne για τις γυναίκες πρόσφυγες. αλλά θα ήθελα να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα Δάφνε που να ωφελήσει και τις γυναίκες πρόσφυγες. Δεν θεωρώ ότι το πρόγραμμα Δάφνε έχει επαρκή κονδύλια ώστε να αφιερώσει κάτι ιδιαίτερα για τις γυναίκες πρόσφυγες. Ως πρόγραμμα κατηγορία 3 και 4 θεωρώ ότι θα μπορούσε να ωφελήσει όμως και τις γυναίκες πρόσφυγες. Συμφωνώ με πολλά από τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε σε ό,τι αφορά τον πολιτικό προσανατολισμό, την πολιτική κατεύθυνση. Και συχνά τα θέματα που αναφέρετε λαμβάνονται υπόψη ήδη και στη νομική βάση για την εκχώρηση των κοντελιών. Ήδη δηλαδή στη φάση αυτή λαμβάνεται υπόψη το συγκεκριμένο θέμα των γυναικών σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το κοινωνικό ταμείο, τα περιφερειακά ταμεία και φυσικά μετά επαφίεται στα κρατημέλη το πώς θα δαπανίσουν τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά, πώς θα τα αφιερώσουν, με ποιο τρόπο θα τα αφιερώσουν στο θέμα των γυναικών. Για το κατά πόσον μπορούμε να έχουν μεγαλύτερες ε, συνεισφορές στον προϋπολογισμό. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε, δεν τυπώθηκε ένα αίτημα το οποίο θεωρώ ότι απέτρεψε ενδεχόμενες μεγαλύτερες συνεισφορές στον προπολογισμό. Το θέμα των σοσιαλδημοκρατών σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό για το Σύμφωνο Σταθερότητας να μην λαμβάνονται υπόψη ε, όλα αυτά τα έκτακτα ή έκτακτες εισφορές σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του ελλείμματος, του δημοσιονομικού ελλείμματος. Να μην ε, ληφθούν υπόψη δηλαδή στον συνυπολογισμό των κριτηριών του Συμφώνου Σταθερότητας. Χάσαμε αυτή την ε, ψηφοφορία Ήταν πιο πολλοί δηλαδή αυτοί που α, καταψήφισαν την πρόταση των χριστιανοδημοκρατών. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία, τι να κάνουμε. Και δεν νομίζω ότι ως Ευρωπαίοι πολιτικοί θα πρέπει να αποτρέψουμε τον, την πιο αποδοτική και αποτελεσματική χρήση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ό,τι ευκαιρία έχουμε για να αυξήσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για να καταστεί πιο αποτελεσματικό. Αυτά. Σα ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην ε, σημερινή μας συζήτηση. Και ελπίζω η γνωμοδότησή μας για τα θέματα ισότητας των φύλων ε, στην εκπόνηση του προϋπολογισμού να ληφθεί με το σωστό τρόπο υπόψη. Τώρα να δούμε το χρονοδιάγραμμα. Η υποβολή της γνωμοδότησης θα γίνει στη συνεδρίασή μας 18 και 19 Απριλίου, προθεσμία για τροπολογίες μέχρι τις 28 Απριλίου 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 13 και 14 Ιουνίου κατά τη συνεδρία της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάθεσης. το οποίο το οποίο είναι, θα έλεγα, δραστηριότητες που προσθέτουν ε, αξία την λειτουργία του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Η Επιτροπή μας πρέπει να υποβάλει την ε, γνωμοδότησή της για το θέμα αυτό και η συγγήτρια είμαι εγώ. Οπότε θα σας κάνω μια παρουσίαση από αυτού. Μέσω της γνωμοδότησης αυτής προσπαθώ να κάνω μια επισκόπηση για τις δραστηριότητες του FC κατά την περίοδο 2007-2014 που πρόσθεσαν προστιθέμενη αξία και ε, στόχευσα τις εξής ε, πλευρές. Πρώτον, οι ωφεληθέντες από το Ταμείο λοιπόν, της Παγκοσμιοποίησης, συγγνώμη, το EAGF, ε, ωφέλησαν 67% τους άνδρες και 37% τους γυναίκες. Και αυτό έχει, έχει να κάνει με τους τομείς απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας με τους, στους οποίους δαπανήθηκαν ε, υπό του Ταμείου και παρά το ότι τα κλώστο υφαντουργικά και οι κοπτοραπτικές δραστηριότητες όπου εργάζονται πάρα πολλές γυναίκες είχαν μεγάλη ανάγκη από χρηματοδότηση από το Ταμείο αυτό. Άλλοι τομεί όπου υπήρχε απασχόληση περισσότερη των ανδρών είχαν ακόμα μεγαλύτερε ανάγκε, για παράδειγμα αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευέ, ε, χαλιβουργία κτλ. Μία άλλη πλευρά επί της οποίας ε, θέλω να επιμείνω είναι ότι οι γυναίκες μπορούν ευκολότερα να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, στην εργασία, αλλά συνήθως αυτή η επανένταξη των γυναικών ε, ε, είναι προσωρινή και επισφαλής. Οι γυναίκες που ψάχνουν για νέα θέση εργασίας ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανακατάρτισης περιορίζονται γιατί πρέπει να φροντίσουν διάφορα μέλη της οικογένειάς τους. Για παράδειγμα δεν έχουν σε ποιον αφήσουν τα παιδιά τους, ε, δεν μπορούν να πληρώσουν βρεφορυμπιακούς σταθμούς, πρέπει να φροντίσουν ηλικιωμένα μέλη της οικογένειάς τους. Οι γυναίκες αυτές δεν έχουν λοιπόν εισόδημα ε, και επειδή προηγουμένως ήταν ε, στην ανεργία δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα για να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιπλέον δαπάνες και αυτό έχει πολύ αρνητική επίπτωση στην επάνω εδώ του στην εργασία. Και κυρίως βεβαίως τι, όπως έλεγα, τις γυναίκες αυτή η κατάσταση. Και ξέρετε ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχει σοβαρή έλλειψη ε, υψηλής ποιότητας ε, και προσιτής ε, βρεφονιπιακής και παιδικής φροντίδας. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί το πλαίσιο λειτουργίας της, του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, ούτως ώστε να στηριχθούν περισσότερο οι γυναίκες που έχουν ε, υποχρεώσει φροντίδας άλλων μελών της οικογένειά του. Μία άλλη πλευρά επί οποία οποίας ε, θέλω να εμείνω, να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα επανένταξη στην εργασία σε τοπικό επίπεδο όπου έχουν προκύψει για παράδειγμα μαζικές απολύσεις για να βοηθήσουν ε, τα άτομα που εργάζονται σε αυτές τις περιοχές ούτως ώστε να μην χρειαστεί να εγκαταλείψουν ε, την ε, περιοχή όπου εργάζονταν προηγουμένως, όπου μένουν για να μην χρειαστεί λοιπόν να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους και αυτό κυρίως αφορά βεβαίως τις γυναίκες οι οποίες είναι πολύ δυσκολότερο να πάνε σε άλλη περιοχή για να βρουν δουλειά ακριβώς επειδή τα παιδιά τους είναι σε ένα σχολείο ή σε κάποιο άλλο ίδρυμα ή αντιμετωπίζουν κάποιους άλλους περιορισμούς αυτές οι γυναίκες δεν μπορούν να πάνε αλλού για να βρουν δουλειά Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω ότι το ποσοστό στήριξης αυτοαπασχολουμένων μέσω πόρων του ταμείου αυτού ήταν μόνο 5%. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να προτείνει μέτρα στα πλαίσια της λειτουργίας του Ταμείου, ε, του ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και κυρίως τη γενική επιχειρηματικότητα. Και τέλος, εφόσον μιλάμε για προστιθέμενη αξία και επίπτωση γενικά του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, θέλω να υπογραμμίσω το ότι φυσικά έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων και προβλημάτων αγοράς εργασίας, ε, ενίσχυσε την κοινωνική συνοχή, βοήθησε στην εξέβρεση νέας εργασίας, Άρα ε, στη δυνατότητα να συμβάλλουν τα άτομα αυτά να παραμείνουν ενεργά, να βοηθήσουν το οικογενειακό εισόδημα και να ε, αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της ανεργίας. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η επανένταξη στην εργασία μέσω στήριξης από το Ταμείο αυτό βοηθάει να αντιμετωπιστεί η ε, εγκατάλειψη κάποιων περιοχών από το εργατικό του δυναμικό και η υποχρεωτική μετανάστευση που όπως ξέρετε μπορεί να προκαλέσει ε, σοβαρά προβλήματα για κάποια κράτη-μέλη, δηλαδή ότι χάνουν ένα σημαντικό τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους. Αυτή είναι μια συνόψιση της γνωμοδότησής μου και να ακούσω τώρα και την ε, δική σας άποψη αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η Μαρία Αρένα. Η Μαρία Ρενά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την έκθεση. Είναι πολύ πλήρης και μας επιτρέπει να δούμε από πλευράς φίλου πώς λειτουργεί ένα ταμείο, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Άρα όταν θέτουμε τα θέματα ισότητας φίλου, το θέμα δεν είναι να υπάρχει χωριστός προϋπολογισμός για την ισότητα του φίλου, αλλά να εξετάζουμε πώς λειτουργούν τα ταμεία για να δούμε αν αντιμετωπίζουν τη διάσταση του φύλου. Νομίζω ότι αναφέρθηκες στο θέμα των κλάδων που φύγονται. Οι κλάδοι, για παράδειγμα, που αναδιαρθρώνονται λόγω της παγκοσμιοποίησης. Πολλοί τέτοιοι κλάδοι είναι κυρίως ε, κλάδοι όπου κυρίως απασχολούνται άντρες, αλλά συχνά είναι θέμα επιλογής που θα χρηματοδοτήσουμε αυτές τις προσαρμογές. Για παράδειγμα, έχουμε πολλές φορές συζητήσει για την ε, ε, υπερπαραγωγή από πλευράς της Κίνας. Βλέπουμε ότι πολλά κράτη ασχολούνται πολύ με τον τομέα της χαλιβουργίας, όπου κυρίως εργάζονται άνδρες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλοί τομείς όπου υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ και περιβαλλοντικό στην Κίνα που δεν ε, λαμβάνουν καθόλου βοήθεια από τα κράτη-μέλη και πολλές φορές και από τα συνδικάτα. Πρέπει λοιπόν να ευαισθητοποιηθούν και τα συνδικάτα για τα θέματα φύλου. Να μην ε, δίνουμε προτεραιότητα μόνο σε τομείς όπου κυρίως ασχολούνται άνδρες. Πρέπει να δούμε ε, πολύ ευρύτερα το θέμα στα κράτη-μέλη. Ε, μπορούν να υπάρξουν άλλοι τομείς. Κλωστεφαντουργία για παράδειγμα έχει αντιμετωπίσει πολύ έντονες αναδιαρθρώσεις όπου δεν είδαμε να υπάρχει βοήθεια από το Ταμείο αυτό να ενημερώσουμε τα κράτη-μέλη, να ευαισθητοποιήσουμε τα συνδικάτα για τα θέματα φύλου όταν υποβάλλουν αιτήματα. Δεύτερον, προσαρμόστηκε ο τρόπος λειτουργίας του Ταμείου αυτού, ούτως ώστε τα άτομα που λάμβαναν βοήθεια να συμπεριλαμβάνουν και τους νέους της περιοχής. Αλλά δυστυχώς οι προτάσεις που γίνονται βλέπουμε ότι όταν γίνεται αναδιάρθρωση σε αρσενικό ας πούμε τομέα κυρίως βοηθάμε την επανεκπαίδευση κυρίως ανδρών. Βεβαίως. Όταν ε, γίνεται μια ευρύτερη προσπάθεια επιμόρφωσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι γυναίκες. Το τρίτον είναι να αξιοποιήσουμε το ταμείο αυτό με τρόπο ιδιαίτερα ενεργητικό. Πολύ συχνά ασχολούμεθα με την αναδιάθρωση ε, μετά τις απολύσεις. Οπότε είναι πολύ αργά. Πρέπει λοιπόν να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Γιατί αλλιώς επειδή δεν υπάρχει ε, νέα οικονομική δραστηριότητα σε αυτή την περιοχή, οι εργαζόμενοι πρέπει να πάνε αλλού. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν αναδιαρθρώσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να βοηθάμε τις γυναίκες να μπορούν και αυτές να βρουν δουλειά στην ίδια περιοχή. Υποστηρίζω πλήρως τις προτάσεις που έκανα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τη Μαρία Αρένα. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Α, με συγχωρείτε. Α, με συγχωρείτε. Κυρία Μέρκελ. Από πλευρά της κυρία Ζαμπόρσκα. Να σας διαβάσω τι έχει να πει. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει η κυρία Ζαμπόρσκα, ω Σκιώδης για την έκθεση αυτή θα ήθελα να κάνω μερικά σύντομα σχόλια σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστώ καταρχάς την κυρία Λεβιτσιούτε για το κείμενό της πολύ χρήσιμο και στηρίζω ιδιαίτερα την άποψή τη. Το ταμείο αυτό και ο κανονισμό για το ταμείο πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τι γυναίκε που έχουν καθήκοντα φροντίδα. Οι περισσότερε γυναίκε αυτέ, η συντριπτική πλειοψηφία είναι εργαζόμενε μητέρε που πρέπει να φροντίζουν και τα παιδιά του. Και οι περισσότερε δεν έχουν καμία δυνατότητα να πάνε αλλού. Δεν μπορούν να αποφεληθούν από πολιτικέ που ενισχύουν την κινητικότητα των εργαζομένων. Οι μητέρε αυτέ ή καλύτερα οι οικογένειες με μικρά παιδιά πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο σε περιπτώσεις απολύσεων. Χρειαζόμαστε περισσότερα επίση στοιχεία για, το, για τους δικαιούχους του ταμείου αυτού. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε σαφέστερα για τι διαφορέ μεταξύ ανδρών και γυναικών και να μην μιλάμε απλώς για προφίλ φίλου. Ο όρο φίλου πρέπει να μα βοηθήσει να συμπεριλάβουμε και ορισμένες ταυτότητες αυτοκαθοριζόμενες. Αλλά εάν θέλουμε να δούμε πόσες γυναίκες έχουν πάρει βοήθεια επειδή έχασαν τη δουλειά τους, ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι κυρίως χάνουν τη δουλειά τους οι γυναίκες και οι οικογένειες με ε, ε, μικρά παιδιά. Ευχαριστώ την κυρία Βιούτε για τη βοήθεια που έχει κάνει για να μας θυμίσει την ύπαρξη της οικογένειας. Ελπίζω να διατηρήσετε αυτές τις διατυπώσεις και να τις επεξεργαστείτε πολύ περισσότερο γιατί νομίζω ότι η ισορροπία μεταξύ εργασία και οικογενειακής ζωή μπορεί να επιτευχθεί μόνο να καταλάβουμε ότι η οικογενειακή ζωή και η φροντίδα των παιδιών είναι τόσο σημαντική για την κοινωνία όσο είναι η απασχόληση και η παραγωγικότητα από πλευρά τη πολιτική μα ομάδα. Συμφωνώ με την κυρία Ελένη Βιτσιούτε ότι πρέπει να στηρίξουμε του αυτοαπασχολούμενους και την επιχειρηματικότητα. Με λίγη βοήθεια και ενθάρρυνση, οι οικογενειακές επιχειρήσει θα μπορούσαν να είναι ιδανική λύση για πολλέ γυναίκε, μητέρε, οικογένειε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Άγκστρομ. Εμένα μου ζητήθηκε η Μόνικα Μάνερ, η σκιώδη των Πρασίνων, να σας μεταφέρω τη γνώμη της. Καταρχάς ευχαριστούμε την εισηγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότησης που αποτελεί καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση για τους πράσινους. Το πιο σημαντικό αίτημα σε αυτή τη γνωμοδότηση θα πρέπει να είναι ότι όσο ε, γίνεται το, η βοήθεια από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης να βοηθά να ωφελεί το ίδιο άνδρες και γυναίκες γιατί δυσανάλογα ε, ε, ε, έχουν πληγεί γυναίκε από την κρίση και θα πρέπει αυτό να αναφέρεται και στη γνωμοδότηση. ειδική μνήμα θα πρέπει να γίνεται στι νέε γυναίκε στην ανεργία. Επίση, πιστεύουμε πω η γνωμοδότηση εστιάζει υπερβολικά στην πτυχή τη μέρημνα τη φροντίδα, που είναι εξαιρετικά βέβαια σημαντικέ για τι γυναίκε αλλά δεν είναι η μόνη πτυχή του Ταμείου που είναι σημαντική για τι γυναίκε. Σα ευχαριστώ. Πόνια λοιπόν, ε, Σλιμ. Ευχαριστώ. Κυρία Σλιμ. Ε, χβάλα ζα ριέτς. Χβάλα οι εισβεστέτελοι Σας ευχαριστώ. Φόντα ζα πριλαγόντμπου γλωμπαλιζάτσι. Στιέλα μπι σάμω δα... Σας ευχαριστώ. Ah. Doprinos ovog fonda na, na odboru za θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια τεχνική πτυχή στην Επιτροπή του Προπολογισμού. Συζητάμε για την ε, κατανομή των κονδυλίων η Πρόεδρος διακόπτει. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τη διερμηνία. Εντάξει τώρα. Okay. Εντάξει, ρυθμίστηκε. Ναι, ρυθμίστηκε. Έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να φτάνουν σε εκείνους που τα χρειάζονται και σε αυτούς που ε, προσπαθούν για να μπορέσουν να έχουν τις νέες δεξιότητες. Οπότε ως Επιτροπή Γυναικών θα πρέπει να φροντίσουμε και να επιστήσουμε την προσοχή στην Κομισιόν ότι αυτή η διαδικασία της ε, κατάργησης της γραφειοκρατίας θα πρέπει να είναι σύντομη, συντομότερη, ώστε τα χρήματα ε, να ε, φτάνουν σε εκείνους που σχεδιάζουν ε, την ε, κατάρτιση των εργαζομένων ώστε να είναι πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν τον λόγο. Νομίζω και θεωρώ πως θα έχουμε και οικοδομητική ε, συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές ώστε να καταλήξουμε σε μια πολύτιμη γνωμοδότηση. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 23η Μαρτίου στις 4 το απόγευμα και η ψηφοφορία θα γίνει στις 18 και 19 Απριλίου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ας συγκεντρωθούμε να περιμένουμε ένα δύο λεπτά και στις 10 ακριβώς θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες σύμφωνα και με την ημερήσια διάταξη.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 ο κ. Γκάιερ. Ήθελα να εκπροσωπήσω μια συνάδελφο σήμερα, αλλά δεν έχω την κάρτα ψηφοφορία μου ακόμα. Μου την φέρνουν και θα ήθελα να ψηφίσω διάθεση ισχύω μέχρι τότε. Yeah. So, uh, uh, Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία μας, λέει η Πρόεδρος. Πρώτη ψηφοφορία εφαρμογή της ε, οδηγίας για την απασχόληση και την ισότητα της κυρίας Σόντροβα. 27, τροπολογία 27, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Άποχες. Θα χρειαστεί να το ελέγξουμε παρακαλώ. Okay. Yeah, yeah. Ah, yeah. Vote is closed. Πέρα τη ψηφοφορία. Μάλλον ε, ξεκινάει η ψηφοφορία και λίγη. Okay. Adopted. It's adopted. Εγκρίνεται. Η 30 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 31 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα χρειαστεί να το ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. δεύτερο τμήμα τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα χρειαστεί ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα χρειαστεί και εδώ ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας αλλάξουμε παρακαλώ και την 52. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 53 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Τροπολογία 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Η τροπολογία 5 έναρξη ψηφοφορίας πέρασα. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Η Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 16. Ε, Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 18. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 19 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η 20 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας ελέγξουμε παρακαλώ τον 25 έναξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 26 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Καλησπέρα. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία. And now it will be three sets for our gender mainstreaming amendment. Και τώρα έχουμε τις τροπολογίες για το gender mainstreaming. Έχουμε την γνωμοδότηση για την Επιτροπή Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά την, ε, τον ιό Ζήκα. Τροπολογία 1. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 1. Έναρξη. Και πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος έναρξη ψηφοφορίας πέρας εγκρίθηκε να σηκώνετε καλύτερα τα χέρια σας αν θέλετε τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τώρα σε ό,τι αφορά την ε, Επιτροπή των Οικολευθεριών και Δικαιωμάτων του Πολίτη. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Η 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Η 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκριθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τροπολογία 3 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Uh, uh, uh, Τώρα το επόμενο θέμα τροπολογίες για την Επιτροπή απασχόληση και κοινωνικών υποθέσεων, η κοινωνική ένταξη και η ένταξη στην αγορά εργασία των προσφύγων. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. πέρα των ψηφοφοριών. Benito Geier. κολέγος, uh, We will continue συνεχίσουμε την ε, συνεδρίασή μας. Τι θέλεις, Άννα, κάτι θέλεις να πεις. Ναι, θέλω σύντομα να παρουσιάσω και να καλωσορίσω κάποιους ε, που θα με συνοδεύουν. IF Metal, δηλαδή ένα συνδικάτο στο το πιο αντροκρατούμενο συνδικάτο ε, αλλά είναι εδώ η συνάδελφος που θα μάθει περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να έρχονται άνθρωποι εδώ, να μαθαίνουν πώς λειτουργεί η Ένωση, τι μπορούν να κάνουν εδώ. Θα με παρακολουθήσει λοιπόν αυτή την εβδομάδα για να μάθει περισσότερα για την Ένωση, για τη λειτουργία της. Σε ευχαριστώ και εγώ σε ευχαριστώ unheard ε, και συμφωνώ πως είναι πολύ σημαντικό να διαδίδονται τα θέματα όσο γίνεται περισσότερο τα θέματα που αφορούν την ισότητα εντός και εκτός της Ένωσης. Να καλωσορίσω λοιπόν τους προσκεκλημένους μας. Και τώρα ας προχωρήσουμε. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες με ιδιαίτερη μνήμα στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Αρμόδιας Επιτροπής του ΟΗΕ. Θα συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης και θα δώσω αμέσως το λόγο στην Ρόζα Εστέβες Φεραγκούτ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Γνωρίζετε ότι από το 2008 έχει συνυπογράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων με Αναπηρία. Είναι το πρώτο νομικό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα το οποίο έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί έτσι τμήμα του νομικού πακέτου και είναι υποχρεωτική εφαρμογή του κατά συνέπεια. Σε αυτήν την ε, αίτηση υπήρχε πρόβλεψη για μια παρακολούθηση και έγινε αυτή η παρακολούθηση και φέτος ο ΙΕ, ο οποίος παρακολουθεί την εφαρμογή, έχει εκδώσει κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες συστάσεις για να δούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά την εφαρμογή αυτή της ε, σύμβασης. Ε, πρόκειται λοιπόν ε, για μια γνωμοδότηση δική μας και αυτά που αναφέρονται ε, στην δική μας νομοδότηση ακολουθούν τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του ΟΗΕ. Όταν, καταρχάς, όταν ε, ε, γίνονται στρατηγικές όπως η στρατηγική για τις ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες ή οι στρατηγικές για τους ανθρώπους με αναπηρία θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το φύλλο πάντοτε. Γιατί η στρατηγική για τον άνδρα και τη γυναίκα δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόβλεψη για την γυναίκα με αναπηρίες. Άρα λοιπόν σε όλες τις στρατηγικές ισότητας φύλου η προοπτική αυτή του φύλου θα πρέπει να είναι παρούσα. Άλλη σύσταση είναι ότι θα πρέπει να γκριθεί και να απεμπλακεί από το Συμβούλιο η οδηγία για τις, κατά των διακρίσεων που εδώ και κάποια χρόνια δεν έχει προχωρήσει. Βρίσκεται στο Συμβούλιο από το 2008 επειδή την μπλοκάρουν κάποιες χώρες. Και κατά τρίτο λόγο υπάρχει το αίτημα, η έκκληση να συνυπογράψουν οι χώρες που δεν το έχουν κάνει ακόμα την σύμβαση της ε, Ισταμπούλ. Ε, γίνεται μία για την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η Σύμβαση θα ήθελε να γίνεται ιδιαίτερη μνήα και για την πρόσβαση των γυναικών κυρίως με αναπηρία στην αγορά εργασίας και ε, ε, πολλοί οργανισμοί και ενώσεις δεν έχουν μπει δεν έχουν προβεί σε αυτές τις προσαρμογές. Επίσης γίνεται αναφορά στην καθολική παιδεία όπου δηλαδή όλοι θα μπορούν να σπουδάσουν, να φοιτήσουν και το, η αναπηρία να μην θεωρείται ως κάτι αρνητικό. Ε, μιλάμε και για τη συνθήκη του Μαρακές που είναι η συνθήκη που θα επιτρέψει στους τυφλούς ή στους δυσκολίες όρασης να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ε, ηλεκτρονικά ε, βιβλία. Ε, και αυτό έχει να κάνει και με το copyright και εκεί υπάρχει μπλοκάρισμα από πλευρά ορισμένων χωρών ε, ε, στο Συμβούλιο για την συνυπογραφή της συνθήκης του Μαρακές. Ετησίως θα πρέπει να, θυμάμαι, να θυμόμαστε ότι το Κοινοβούλιο μας είναι μέρος αυτού του πλαισίου εποπτείας, δεν θα πρέπει αυτό να το ξεχνάμε και για, είμαστε υπεύθυνοι και για ό,τι έχει να κάνει με το συντονισμό έχουμε να κάνουμε για την την αναπηρία. Το θέμα της αναπηρίας είναι οριζόντιο, δεν είναι μόνο η γυναίκα, είναι η γυναίκα, είναι οι μεταφορές, είναι η παιδεία, είναι η ψηφιακή εποχή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε αυτές τις οριζό, τους οριζόντιους μηχανισμούς. Και έπειτα, πολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι ακόμα ένας πολύ σημαντικός άξονας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με τις τροπολογίες σας θα βελτιώσουμε το κείμενο. Είμαι εισηγήτρια και σε άλλες επιτροπές όπως στην Επιτροπή Πέτη είμαι Σκιώδη, στη Γιούρη επίσης. Γι' αυτό και θα πρέπει πιστεύω να επηρεάσουμε την τελική έκθεση όσο γίνεται περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Φερακούτ. Ιάννα Γκέρτ. Σας ευχαριστώ. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελε να ευχαριστήσει την εισηγητρία. Γιατί πιστεύουμε ότι γενικά η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή. Και σίγουρα συμφωνώ και με την εισηγητρία ότι είναι πραγματικά ε, τρομερό το γεγονός ότι η νομοθεσία αυτή κατά τον διακρίσεων δεν έχει εφαρμοστεί. Ε, ε, παρά το γεγονός ότι συζητιέται επί τόσα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η νομοθεσία για τα άτομα αυτά με αναπηρία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να ασκούμε πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Και σε ό,τι αφορά την προς υπογραφή της συνθήκης. Τώρα θα ήθελα να κάνω και κάποια σχόλια. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόταση, όπου για παράδειγμα χρησιμοποιείται ε, σεξουαλική εκμετάλλευση. Πολλά άτομα με αναπηρία είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Όχι μόνο θύματα βίας, αλλά και σεξουαλικής βίας συγκεκριμένα. Θα καταθέσω λοιπόν μια σχετική τροπολογία. Φυσικά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να βοηθεί, βοηθάτε Φυσικά λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη και όσο ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη να εξετάζουμε τα θέματα λοιπόν της εφαρμογής της νομοθεσίας, της σύμβασης της Ισταμπούλ, της συνθήκης της Μαρακές και των σχετικών ζητημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λέκη Πρόεδρος. Veľmi pekne. Ε, Σας ευχαριστώ και εγώ θα είμαι σύντομη. Θα, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το εξαιρετικό της κείμενο. Δεν υπάρχει πολλή χώρο και είναι δύσκολο να πει κανεί όσα θέλει στον περιορισμένο αυτό χρόνο. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε με τροπολογίε αυτή την έκθεση. Ε, θέλω να αναφερθούμε και στις ε, ε, εκπαιδευτικές απαιτήσει και δυνατότητες και μέσω της παιδείας είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, διακρίσεις έναντι των ε, ανθρώπων με αναπηρία. Ταυτόχρονα όμως είναι απαραίτητο να μιλήσουμε για την βία που ασκείται κατά των ανθρώπων με αναπηρία. Αυτές, αυτή η βία δεν ασκείται μόνο μέσα στα ιδρύματα αλλά και ε, στο οικιακό περιβάλλον, στις μέσα, είναι ενδοοικογενειακή βία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους και αυτά τα θύματα. Υπάρχει μια ακόμα αρχή που θα ήθελα να συμπεριληφθεί σε αυτό το κείμενο. Η ιδέα δηλαδή του να είναι εγγυημένη εγγυημένο το μεγαλύτερο όφελο στο συμφέρον μάλλον του ανηλίκου, του παιδιού κάθε φορά. Γιατί υπάρχουν και τα παιδιά με αναπηρία που πολύ συχνά θεωρούνται βάρος, υπόκειται σε διακρίσεις, αν και θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν και να ενταχθούν και σε στάνταρ σχολεία και πολλές φορές μάλιστα αντί να τα κρατήσουν οι οικογένειε τους, τα τοποθετούν σε ιδρύματα. Το θέμα είναι πώς θα βοηθήσουμε τις οικογένειες να τα κρατήσουν τα παιδιά του σπίτια τους, να ευαισθητοποιήσουμε τα κρατημέλη ώστε να εγγυηθούν τη βοήθεια για τις οικογένειες με τέτοια παιδιά ή, ε, ή για τα, τους και τα ιδρύματα που βοηθούν τις οικογένειες με τη σειρά τους χωρίς να διαλυθούν ε, γιατί πολύ συχνά οι οικογένειες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ε, όταν έχουν παιδιά με αναπηρία ε, και δυστυχώς το τέλος δεν είναι πάντοτε αίσιο. Αυτά λοιπόν και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ και τώρα η κυρία Χιμένες ζήτησε το λόγο. Ε, ε, ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την εργασία της για τα άτομα με αναπηρίες, όχι μόνο εδώ στην Επιτροπή μας. Όπως σωστά είπε, είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους τομείς πολιτικής. Αφορά όλη, όλες τις πλευρές της ζωής. Την ευχαριστώ για την εργασία της, για ε, τον αγώνα που έχει κάνει για τα άτομα με αναπηρία. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η κύρια ή τουλάχιστον από τις κύριες δραστηριότητές της και τώρα στο Κοινοβούλιο και πριν. Είναι πολύ πλήρης αυτή η έκθεση. Δεν έχουμε πολύ χώρο βέβαια, οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε όλα όσα θέλαμε. Αλλά συμφωνώ και με την προηγούμενη ομιλήτρια που έθεσε το θέμα των ανηλίκων και ιδίως το θέμα των κοριτσιών με αναπηρίες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα. Έχω μιλήσει με γυναίκες με αναπηρία. Σε πολλές χώρες δεν λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματά τους. Όταν παντρεύονται, για παράδειγμα, όταν έχουν συναισθηματικές σχέσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αναπηρίες τους. Το θέμα δεν είναι ότι έχουν διανοητική αναπηρία. Είναι δύσκολο να τα βγάλουν πέρα γιατί η νομοθεσία της κάθε χώρας είναι διαφορετική, είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Πρέπει να επιμείνουμε και στο οικονομικό θέμα γιατί πολλές φορές τα άτομα με αναπηρίες είναι και άτομα φτωχά. Χρειάζονται λοιπόν βοήθεια. δεν πρέπει να παρετούμεθα των δυνατοτήτων που έχουμε να τους βοηθήσουμε, να αρνούμεθα τις ευθύνες μας. Πρέπει όλοι να υπογράψουν την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Γιατί μόνο έτσι αισθάνονται ότι έχουν ρόλο στην κοινωνία και τα άτομα αυτά. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την έκθεση, να δούμε τι άλλο μπορούμε να πούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι ήδη πολύ καλή και πολύ πλήρη και πλήρης αυτή η έκθεση και την ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Χιμένεθ Μπεσερίλ. Και τώρα από πλευρά τη Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή σας για τις σκέψεις και συστάσεις που περιέχονται σε αυτή τη γνωμοδότηση που βοηθούν πολύ στην εφαρμογή της σύμβασης. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εφαρμοστούν οι καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και σας διαβεβαιούμε ότι αποδίδουμε την απαραίτητη σημασία να ενισχυθεί η οπτική φύλου κατά την εφαρμογή των δράσεων αυτών όπως υπογραμμίσατε και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Η κυρία Σταράς Φεραγκούτ. Φεραγκούτ. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Ευχαριστώ και για την παρουσία της Επιτροπής που ήταν ε, ε, στήριγμα όταν ε, θέλησα να εργαστώ για το θέμα αυτό η ψηφιακή πρόσβαση, το δικαίωμα πρόσβαση στην εργασία, η απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς, συγγνώμη, εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς Όλα αυτά βοηθούν και τις γυναίκες με αναπηρίες. Αυτή είναι η πρόκληση. Να τα επιτύχουμε όλα αυτά και για την Επιτροπή μας. Η γυναίκα με αναπηρίες, όπως ξέρετε, έχει ένα διπλό μειονέκτημα. Έχει την αναπηρία της και έχει και την κατάστασή της ως γυναίκα. Όλοι συμφωνούμε με τη σύμβαση βεβαίως αλλά πρέπει να δούμε και τι έχουν κάνει τα κράτη-μέλη και η ίδια η Ένωση για την εφαρμογή αυτής της ε, σύμβασης. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει πολύ περισσότερα. Γιατί από το 2008 έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια. Και ούτε κάνει στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες δεν έχει ένα χωριστό τμήμα για τις γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να μας χρησιμεύσουν αυτές οι καταληκτικές παρατηρήσεις για να αλλάξουμε τον τρόπο αντιμετώπισης γιατί αυτή η σύμβαση λέει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί όλη η ευρωπαϊκή νομοθεσία για να προσαρμοστεί στη σύμβαση. Και αυτά μας τα έχει πει εδώ και 8 χρόνια, αλλά δεν έχει γίνει αυτό. Άρα η δουλειά μας, ε, η δουλειά μας πρέπει να συνεχιστεί τροπολογίες μέχρι τις 26 Μαρτίου, όπως σωστά είπε η σύντροφός μου εδώ. Βεβαίως με αυτήν την γνωμοδότηση μόνο ένα παραπάνω μπορούμε να κάνουμε αλλά είμαι σίγουροι ότι με τι τροπολογίε όντω θα συμπληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα μόνο να σα υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών είναι η 29η Μαρτίου στις 3 το απόγευμα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Μια και προχωρήσαμε γρήγορα. Σήμερα λοιπόν στην Επιτροπή μας έχουμε μια αντιπροσωπεία γυναικών βουλευτών από τη Βουλή της Μολδαβίας. για την αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου της Μολδαβίας, η οποία είναι και επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτής. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων για, την, για το ρόλο των γυναικών στην πολιτική. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερως όταν πρόκειται για όμορφε χώρε Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η πτυχή αυτή. Και είναι σημαντικός ε, ο διάλογος αυτός και πολύ επίκαιρος, μιας και η Επιτροπή μας καταρτίζει μια έκθεση για τα δικαιώματα των γυναικών στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και στις άλλες γειτονικές χώρες. Θα θέλαμε ως τούτου λοιπόν να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις για την κατάσταση των γυναικών, για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε για να εφαρμόσουμε αυτή την αρχή της ισότητας των φίλων σε όλα τα πεδία. Είναι σημαντική λοιπόν η ανταλλαγή αυτή αντιπόψεων. Και χαιρόμαστε που μας επισκέπτεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία Λιλιάνα Μολιχοβίτση, η οποία είναι αντιπρόεδρος της ε, Μολταβικής Βουλής. Έχετε το λόγο. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρευρεθούμε εδώ σήμερα σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής και να παρουσιάσουμε και τις δικές μας πληροφορίες σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των ε, ευρωπαϊκών πολιτικών που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ και εκπροσωπούμε το Μολδαβικό Κοινοβούλιο. Επτά γυναίκες λοιπόν, μέλη του συντονιστικού, α, της Συντονιστικής Επιτροπής για την ειρήνη στο κοινοβουλίο μας. Μας πήρε πάρα πολύ καιρό η δημιουργία αυτής της Επιτροπής στο κοινοβουλίο μας και για πρώτη φορά σε 25 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας μας καταλήξαμε σε μια κοινή θέση σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και την κοινή διατύπωση απόψεων από όλο το πολιτικό φάσμα συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια θέματα τα οποία μας ενώνουν και θα πρέπει να προαγάγουμε ζητήματα τα οποία θα βελτιώσουν τη ζωή των γυναικών στη δημοκρατία της Μολδαβίας. Σήμερα θα πρέπει να συζητήσουμε, είπατε, την πολιτική συμμετοχή των γυναικών, αλλά δεν μπορώ να περιοριστώ στο θέμα αυτό, γιατί η πολιτική συμμετοχή των γυναικών προϋποθέτει ότι θα έχουν πληθεί και κάποια άλλα προβλήματα, προκειμένου να είναι πιο δεσμευμένε. πιο σίγουρες οι γυναίκες για τις εξουσίες που έχουν, για τις δυνάμεις που έχουν και για την δυνατότητα επιρροής της πολιτικής ζωής στην περιοχή που μένουν, που ζουν. Σήμερα είμαι εδώ με την κυρία Μπούλικα, η οποία εκπροσωπεί την Δημοκρατικό Κόμμα και είναι πρόεδρος της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και για την πολιτική εξωτερικών υποθέσεων, η κυρία η οποία εκπροσωπεί του φιλελεύθερου μέλο της Επιτροπής εκπαίδευση Αθλητισμού και Μέσων ενημέρωση, η κυρία Αλίνα Ζώτα, η οποία εκπροσωπεί τους φιλελεύθερου και είναι μέλος της Επιτροπής για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και για την Ευρωπαϊκή Ενωπήση. Η κυρία Μπάλμο είναι μη εγγεγραμμένο μέλος του Κοινοβουλίου, μέλο τη Επιτροπή για την Κοινωνική Προστασία και έχουμε και την κυρία Ντομέτη, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής για την Κοινωνική Προστασία και την Υγεία. Η κυρία Ντολίντσα είναι εκπρόσωπος των σοσιαλιστών, μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου μας. Και γιατί σας παρουσιάζω λοιπόν τις συναδέλφους, για να σας ε, καταδείξω ότι εκπροσωπούμε πραγματικά όλο το πολιτικό φάσμα της Μολδαβίας, ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις ε, μεταξύ των κομμάτων. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων και του Κοινοβουλίου υποστηρίζει την, ε, το δημοκρατικό δρόμο της ευρωπαϊκής διάστασης. Κάποιοι ήταν κατά της ευρωπαϊκής διάστασης της Μολδαβίας, αλλά συμμετείχαν ε, στι αντιπροσωπείε μα και σήμερα κατανοούν ότι η μοναδική ευκαιρία για την εξέλιξη και την πρόοδο στη χώρα μας είναι η δυνατή, στεναρή εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνέχιση εφαρμογή στη χώρα μας των ευρωπαϊκών αξιών. Θα πω εν συντομία δύο λόγια για την πλατφόρμα μας. θεωρούμε ότι επί 25 χρόνια στη Μολδαβία αγωνιζόμαστε για να συμμετοχούν πιο πολλέ γυναίκε στο Κοινοβούλιο, για να επηρεάζουμε τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο. Εξακολουθούμε να αποτελούμε ένα 22% των συνολικών βουλευτών. Τα τελευταία δύο χρόνια εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να προωθήσουμε την τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις για τη συμμετοχή των γυναικών. Και σήμερα στο Κοινοβούλιο ε, περνάει από δεύτερη ανάγνωση ένα νομοσχέδιο το οποίο προτείνει ακριβώς τέτοιες τροπολογίες στην Εθνική Νομοθεσία. Η πλατφόρμα μας διαπραγματεύεται με τα πολιτικά κόμματα το πώς θα ψηφίσουν, γιατί έχουμε κάνει κάποιες τροπολογίες ε, προς την πρόταση αυτή σε ό,τι αφορά την εισαγωγή υποχρεωτικών ποσοστώσεων ύψους 40% στο Κοινοβούλιο κάποιοι ζητούν 30%, 35%, 50%. Διεξαγάγουμε λοιπόν αναλύσεις σχετικά με το θέμα αυτό και προτείνουμε μία ποσόστοση την οποία θα υποστηρίξει τελικά η πλειοψηφία των βουλευτών προκειμένου να συμπεριληφθεί αυτή η ποσόστοση στην νομοθεσία. Γιατί οι αλλαγές αυτές θεωρούμε ότι οι αλλαγές που επιθυμούμε να γίνουν δεν θα καταφέρουμε να τις πετύχουμε χωρίς υποχρεωτικές ποσοστώσεις. Ίσως μετά από με την πάροδο του χρόνου αυτό να καταστεί κάτι κανονικό και αυτονόητο και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να βγει από την νομοθεσία μετά. Το θέμα δεν είναι να υπάρχει ποσόστοση καθε αυτή. Το θέμα είναι πώ θα μπουν και οι γυναίκε ε, στι λίστε των πολιτικών κομμάτων. Γιατί έχουμε πολιτικά κόμματα σήμερα που έχουν πάνω από 30% γυναίκες στις λίστες τους. Αλλά οι γυναίκες δεν μπαίνουν σε θέσεις που να έχουν ευκαιρία να μπουν στο κοινοβούλιο. Είναι στο δεύτερο τμήμα, για παράδειγμα, της λίστας. Αυτό φυσικά δεν βοηθάει τις γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν ένας στόχος της πλατφόρμα μας είναι να συνεργαστούμε με βουλευτές από διάφορα πολιτικά κόμματα για να καταφέρουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ψηφιστεί το έγγραφο αυτό. Επίσης, ένας άλλος στόχος της πλατφόρμα μας είναι να επηρεάσουμε και να συμβάλλουμε στην αλλαγή νοοτροπίας του κόσμου. Πώς θα εκλεχθούν πιο πολλές γυναίκες στο κοινοβούλιο αν η κοινωνία θεωρεί ακόμα ότι η θέση τη γυναίκας είναι στην κουζίνα και όχι στη λήψη αποφάσεων. Έχουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά μελέτε και έρευνες που έγιναν στην Δημοκρατία της Μολδαβίας και τα στοιχεία λοιπόν αυτά καταδεικνύουν ότι περίπου 79% των ερωτηθέντων στην έρευνα αυτή θεωρούν ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα και όχι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό το τμήμα λοιπόν του πληθυσμού εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν είναι σε θέση, δεν είναι έτοιμες να συναγωνιστούν για υψηλόβαθμες θέσεις. Ακόμα και αν παρά το γεγονός ότι και στην Μολδαβία έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά εκπαιδευμένων γυναικών με πανεπιστημιακά πτυχία. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι η πλειοψηφία των αποφύτων από τα πανεπιστήμια είναι γυναίκες. Όταν βλέπουμε όμως τι γίνεται στις θέσεις απασχόλησης, τα πράγματα αντιστρέφονται. Εδώ τίθεται και ένα θέμα αντίληψη και κατανόησης. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι καθήκον της πλατφόρμας μας, να έχουμε καλή επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών για τέτοια ζητήματα και θέλουμε να δώσουμε πιο πολύ ορατότητα στις γυναίκες από το Κοινοβούλιο, στις βουλευτές, ευθύνες. Να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των γυναικών στην Μολδαβία, προκειμένου να αλλάξει και αυτή η νοοτροπία, αυτή η αντίληψη του κόσμου. Σημειώθηκε κάποια μικρή αλλαγή. Σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2010 και αυτό χάρη σε διάφορες ε, δραστηριότητες που αναλάβαμε. Το 2010 λοιπόν, για παράδειγμα, περίπου 67% των ερωτηθέντων θεωρούσαν ότι μόνο οι γυναίκες μπορούσαν να θρέψουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά. Ότι οι άντρες δεν μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά. Δεν έχουν την ικανότητα, δεν έχουν δυνατότητα. 67% Σήμερα 80% του πληθυσμού θεωρούν ότι οι άντρε έχουν την ε, δυνατότητα να μεγαλώσουν ένα παιδί. Και αυτή η αλλαγή λοιπόν οφείλεται και στις αλλαγές της νομοθετικές από πλευρά του Κοινοβουλίου δώσουμε μεγάλη δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωση. Για να δείξουμε ότι και η γονική άδεια, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από τις γυναίκες, αλλά και από τους άνδρες. Και ότι και οι άνδρες θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες για να συμμετάσχουν στην ανατροφή των παιδιών. Αυτό επέφερε αλλαγέ λοιπόν στην ε, νοοτροπία του κόσμου. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να προβληθούν. Να προβληθούν τέτοια μηνύματα προ το κοινό. Μία άλλη δραστηριότητα που σχεδιάζουμε από πλευρά τη πλατφόρμα το Μάρτιο του 2016 μέχρι το 2018 είναι μία δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τι γυναίκε γιατί έχουμε πραγματικά κουραστήρια να συζητάμε τα προβλήματα των γυναικών χωρίς αποτελέσματα. Και βλέπω ότι αυτό συμβαίνει και σε διεθνή συνεδρία σε πολλές περιπτώσεις. Ε, εντάξει, μαζευόμαστε, συζητάμε τα προβλήματα και τελικά οι κυβερνήσεις, οι εθνικές δεν ε, λαμβάνουν μέτρα. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει η προσέγγιση και στο φόρουμ μας, γιατί γεωργανώνονται διάφορες ε, εκδηλώσεις και στη χώρα μας. Για φέτος Διοργανώνουμε λοιπόν ε, στο φόρουμ εννέα ομάδες εργασίας και αποφασίσαμε να δημιουργηθούν αυτές οι ομάδες εργασίας για προβλήματα, για ζητήματα τα οποία απασχολούν διάφορες ομάδες γυναικών στη Μολδαβία. Έχουμε για παράδειγμα τις γυναίκες με HIV, γυναίκες επιχειρηματίες, γυναίκες δημοτικές σύμβουλοι κοιτάμε τι προβλήματα συγκεκριμένα αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές και πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Έχουμε μία ομάδα για την ενσωμάτωση στην διεθνή ε, αγορά εργασίας για γυναίκες που έρχονται από το εξωτερικό. Ξέρετε ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό ε, γυναικών που εργάζονται στο εξωτερικό. Και σε ό,τι αφορά την ε, διασπορά της Μολδαβίας, διαπιστώνουμε ότι σε πολλές περιπτώσει θέλουν να επιστρέψουν, αλλά αντιμετωπίσουν πρόβλημα για να μπουν στην αγορά εργασία, για να μπουν τα παιδιά τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της Μολδαβίας. Αποφασίσαμε λοιπόν να αφαιρεθεί μια ομάδα εργασία σε αυτέ τι γυναίκε, να συζητήσει τα θέματα αυτά και τι δράσει που θα χρειαστεί να προωθήσει και το Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση. Και η ιδέα λοιπόν ε, του φόρουμ αυτού είναι να προσκληθούν όλοι οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο σήμερα προκειμένου να συνομιλήσουν με εκπροσώπους από όλες τις ομάδες εργασίας. 40 λεπτά θα έχει στη διάθεση του κάθε επικεφαλής ε, κόμματος, κάθε πρόεδρος κόμματος, με κάθε ομάδα εργασίας και τελικά θα πρέπει να καταλήξουν στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τι θα κάνουν για χρονική περίοδο ενός έτους για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της κάθε ομάδας εργασίας. Σε ένα έτος λοιπόν θα ξαναδιοργανωθεί ένα φόρουμ, θα ξαναπροσκληθούν οι συγκεκριμένοι πρόεδροι κομμάτων για να πούν στο κοινό τι έκαναν στο κοινοβούλιο για να υποστηρίξουν τις γυναίκες και πώς συγκεκριμένα συνέβαλαν στην επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Θέλουμε οι πολιτικοί να συμμετέχουν και να αισθάνονται πιο υπεύθυνοι για θέματα γυναικών. Έχουμε και προγράμματα για να δίνουμε συμβουλές, μέντορες, ούτως ώστε να μαθαίνουν και οι νέες τι κάνουμε εμείς στο Κοινοβούλιο και για να γίνονται πιο μαχητικές, να συμμετέχουν στην ομάδα μας, στην ομάδα γυναικών που θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή για το λαό της Μολδαβίας. Ευχαριστώ πολύ και με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Λιλιάνα Παλεχόβιτς. για αυτήν την παρουσίαση που μας κάνατε της κατάστασης των γυναικών στη χώρα σας, την Δημοκρατία της Μολδαβίας. Και τώρα παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα η κυρία Νταντσίλα. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα προσεκτικά αυτά που μας είπαν οι συνάδελφοι από την Μολδαβία και νομίζω ότι περισσότεροι καταλαβαίνουμε πολύ καλά, μπορούμε να ταυτιστούμε με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν γιατί η Επιτροπή μας και γενικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει ζητήσει για το πώς θα προωθηθούν οι γυναίκες όχι μόνο στην πολιτική, στην επιστήμη, την έρευνα και άλλους τομείς δραστηριότητας όπου αντιμετωπίζουμε την ε, αόρατη, τη γυάλινη όπως λέμε οροφή όταν προσπαθούμε να ανέβουμε. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις γυναίκες μέσω ποσοστώσεων και άλλων μέτρων και συνεργασίας όλων των πλευρών. Γιατί το θέμα δεν είναι κάτι που αφορά κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Όλα τα κόμματα λένε ότι θέλουν να στηρίξουν τις γυναίκες, αλλά μετά ε, στην πράξη όλοι λένε ότι υπάρχουν πολλές δυσχέρειες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ενότητα μεταξύ όλων των κομμάτων. Και πριν προσπαθήσουμε να αναλάβουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες, πριν προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε κανόνες, πρέπει πρώτα απ' όλα, σε άλλους δηλαδή, Πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση και στο εσωτερικό των κομμάτων μας. Εγώ είμαι πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών Γυναικών στη Ρουμανία και υπέβαλα μια πρόταση απόφασης το καλοκαίρι όπου έλεγα ότι τουλάχιστον 30% ποσοστός θα πρέπει να υπάρξουν στην πολιτική. Και όταν λέω πολιτική δεν αναφέρομαι μόνο στο Κοινοβούλιο, αναφέρομαι και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Διότι Μια τέτοια απόφαση πραγματικά θα βοηθούσε την κατάσταση των γυναικών. Έγινε δεκτή από το κόμμα η απόφασή μου, αλλά και οι γυναίκες ε, σε άλλα πολιτικά κόμματα επέβαλαν ε, παραπλήσεις αποφάσεις και ελπίζω ότι τώρα θα μπορέσουμε να υποβάλουμε και μία νομοθετική πρόταση σε ενωσιακό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες στην πολιτική να το δούμε αυτό από δύο απόψεις. Πρώτα απ' όλα οι γυναίκες είναι μαχητικές, είναι θαραλές. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουν το βήμα, να εμπλακούν στην πολιτική γιατί πολλές φορές διστάζουν να εμπλακούν σε πολιτική δραστηριότητα και επίσης θα πρέπει να είναι ενωμένες οι γυναίκες σε όλα τα πολιτικά κόμματα Ούτω ώστε να αυξηθεί λοιπόν το ποσοστό συμμετοχή του ε, στι γυναίκε όπου είναι, ε, χώρες που είναι ακόμη χαμηλό. Πιστεύω λοιπόν ότι και για τη Ρουμανία, για τη Μολδαβία, για τη Βουλγαρία αλλά και για άλλε χώρε οι ποσοστώσει είναι η μόνη λύση. Η μόνη λύση που μα έχει απομείνει για να επιβάλλουμε την παρουσία γυναικών στην πολιτική. Έτσι θα έχουν πρόσβαση στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και αυτό πιστεύω ότι θα βελτιώσει τη ζωή πολλών γυναικών είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε εργάζονται στην Ήπεθρο, γιατί νομίζω ότι οι γυναίκες καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες γυναίκες, ε, τις διακρίσεις που υφίστανται και στην σταδιοδρομία τους και στην οικογενική τους ζωή, τις δυσχέρειες και ε, για να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι υπέρ του στόχου της ένταξης ε, της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι όλες οι γυναίκες ε, πρέπει να το στηρίξουν, γιατί αυτό θα βοηθήσει την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ε, πρόθεση των θεμελιωδών αξιών που θέλουν και οι γυναίκες και για τους εαυτούς τους και για τα παιδιά τους. Πολλά μπορούμε να πούμε ακόμη, αλλά πιστεύω ότι η παρουσία των συναδέλφων μας από την Μολδαβία εδώ και ο τρόπος με τον οποίο προωθούν τα συμφέροντα των γυναικών είναι αυτός που και εμείς ε, προσπαθούμε να προωθήσουμε για τις γυναίκες στις δικές μας χώρες και πιστεύω ότι από κοινού μέσω καλής συνεργασίας μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα που είναι σημαντικά και για μας και για τις γυναίκες που περιμένουν εμείς να μην τις στηρίζουμε μόνο στα λόγια αλλά στην πράξη με συγκεκριμένα μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρξουν και νομοθετικά μέτρα και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και σας ευχόμεθα κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ντανσίλα και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, κυρία Κουζλόφικα. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να, ε, καταρχάς να συγχαρώ θερμά τους, ε, τις συναδέλφους από τη Μολδαβία. Ε, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ και μάλιστα ήθελα να σας συγχαρώ για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχάς ήρθατε εδώ αντιπροσωπεύοντας διάφορα πολιτικά κόμματα. Είστε καλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει ελπίδα για την ε, Μολδαβία και το λέω αυτό γιατί πρόσφατα έγιναν διάφορες συζητήσεις που χρωματίστηκαν από απογοήτευση για τη χώρα σας. Είναι σημαντικό λοιπόν που είστε σήμερα εδώ γιατί δείχνετε πόσο σημαντικές είναι οι γυναίκες για την πολιτική της ε, χώρας αλλά και αλλά ταυτόχρονα και ότι βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει μια κοινή προσπάθεια που ξεπερνά τα σύνορα των διαφορών πολιτικών κομμάτων. Πολύ σημαντικό που είστε λοιπόν στο Κοινοβούλιο της χώρας σας και που επισήμως αντιπροσωπεύετε τις γυναίκες, γιατί πολύ συχνά οι γυναίκες ικανοποιούνται με άτυπες δυνατότητες να κάνουν ε, θετικά και δράσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό που εσείς αγωνίζεστε επίσημα ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των ε, πολιτών και του γυναικείου κομματιού της. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η ζωντανή ανάμειξη θα σας επιτρέψει να προσελκύσετε περισσότερες γυναίκες στην πολιτική γιατί είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι μας. Θυμάμαι στη Πολωνία η οι Πολωνέζες φεμινίστρες συνήθιζαν να έρχονται σε επαφή με βουλευτές του Κοινοβουλίου. Κάποιες φορές είχαν συναντήσει τον Πρωθυπουργό και ζητούσαν το gender mainstreaming. Τόνιζαν ότι οι γυναίκες όχι, δεν θέλουν πια να κάνουν παιδιά, όχι γιατί δεν έχουν όρεξη, αλλά λόγω των εμποδίων, λόγω της έλλειψης ε, ε, ε, εικόνα για τις οικογένειες και το γεγονός ότι ε, δηλαδή οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ορθότερες οικογενειακές πολιτικές και το γεγονός ότι είστε εδώ είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά ποσοστώσεις για τις γυναίκες, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερη και η μόνη λύση. Ε, ας πούμε, αν σκεφτεί κανείς τις λύσεις που έχει εφαρμόσει η Σουηδία και άλλες χώρες είναι πολύ καλύτερες. Όμως το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να είναι πολύ ε, ακριβές οι λύσεις αυτές, ενώ η ποσοστός είναι ένα σχετικά φθηνός τρόπος ώστε να υπάρξει μια αλλαγή και να επιστηθεί η προσοχή της κοινωνίας στο γυναικεία προβλήματα. Αξίζει λοιπόν να το προσπαθήσει κανείς γιατί έτσι μπορεί να κάνει πολλά σε σχετικά σύντομη χρονική περίοδο. Τέλος, να σας πω ότι έχουμε σύνοδο στον ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε το πρώτο φόρουμ γυναικών ε, που θα διοργανωθεί παράλληλα θα συμμετέχουν ε, γυναίκες από τα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής ε, Γειτονίας. Είστε ευπρόσδεκτες, θα βρείτε τις προσκλήσεις βέβαια και στα mail σας. Παρακαλώ λοιπόν αν θέλετε να έρθετε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κοσλοφκέιβ. Και τώρα η κυρία Ρέντκε. Θέλω να σας καλωσορίσω θερμά. <coughs> Συγγνώμη που δεν σας κοιτάω, Έχω αλλά είναι επειδή κάθομαι σε αυτή τη θέση. Όταν μιλούσατε για την κατάσταση των γυναικών στην Μολδάβα, μου θύμισε την κατάσταση ε, των γυναικών σε άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Όταν, ας πούμε, μιλήσατε για τις προκλήσεις όσον αφορά την ε, συμμετοχή στην πολιτική ζωή, αλλά και τις προκλήσεις στην ισορροπία της οικογενειακής με την εργασιακή ζωή, παρόμοιους αγώνες δίνουμε και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ανταλλάσσουμε ε, τις απόψεις μας. Και θέλω να τονίσω τρία πράγματα που συζητάμε εδώ, σε αυτή την Επιτροπή, τρεις νομοθετικές προτάσεις που βρίσκονται επιτάπητος, που θα προταθούν σύντομα, όπου έχουμε... Έχετε ήδη αναφέρει τα θέματα. Το ένα είναι τα, οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, που δεν εξετάζουμε μόνο το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στα πολιτικά όργανα, αλλά και στην συμμετοχή των γυναικών στην λήψη οικονομικών αποφάσεων. Γίνονται τέτοιες συζητήσεις και σε εσά, γιατί πολλοί, από την εξουσία στις, στις κοινωνίες μας ε, βρίσκεται στις, ε, στα οικονομικά περιβάλλοντα και εκεί που λαμβάνονται οικονομικές αποφάσεις. Ε, άλλο θέμα είναι η αναθεώρηση της οδηγίας για την ε, άδεια μητρότητας εδώ στο Κοινοβούλιο και κάτι που θέλει οπωσδήποτε η Κομισιόν να προσθέσει είναι η άδεια πατρότητας. Εσείς μας δώσατε ενδιαφέροντα στοιχεία για το κατά πόσο και οι άντρες ε, φροντίζουν τα παιδιά ή μεγαλώνουν τα παιδιά πιστεύετε ότι, μάλλον συζητάτε αυτό το θέμα, γιατί πιστεύουμε πως πρέπει οι άντρες να αναμενύονται περισσότερο στην υπόθεση της ανατροφής των παιδιών, αλλά και στις ε, ιδρύματα φροντίδας για τα παιδιά. Μετά, έχουμε το θέμα της ε, ίσης αμοιβής. Έχουμε Ας πούμε στη Γερμανία η διαφορά είναι 22% της αμοιβή για ίση εργασία Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλο το πρόβλημα, οδηγεί και σε διαφορά μεγάλη και στις συντάξεις. Έχουμε πρόβλημα φτώχεια στις γυναίκες μεγαλύτερο και είναι θέματα στα οποία νομίζω πρέπει να δουλέψουμε για να έχουμε μια πιο <coughs> δίκαιη κοινωνία. Κάτι ακόμα που το αναφέρατε, λέει, μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες περικές λεπτομέρειες. Είπατε ότι συνεργάζεστε και με τα κόμματα. Πιστεύω και εγώ ότι τα πολιτικά κόμματα παίζουν κρίσιμο ρόλο για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Εσείς αναφέρατε προγράμματα ε, συνοδών ή νονών. Έχετε άλλο είδους συστήματα. Αναφέρατε ότι οι γυναίκες έχουν μπει σε εκλογικούς καταλόγους σε θέσεις όπου δεν πρόκειται ποτέ να εκλεγούν και εμείς το έχουμε δει και το ζούμε αυτό. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά λοιπόν για την συνειδητοποίηση και μέσα στα ίδια τα πολιτικά κόμματα. Ίσως μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ λέει Πρόεδρος. κυρία Žao mi što nisam Σας ευχαριστώ. Λυπάμαι που δεν συμμετείχα εξ αρχή στη συζήτηση αυτή, αλλά θα ήθελα να πάρω και εγώ το λόγο, γιατί όσο πιο πολλά ακούω, τόσο πιο πολύ μου αρέσει η ιδέα της ποσόστοσης, γιατί αν και δεν θα σας αρέσει αυτό που θα πω, Θεωρώ ότι οι ποσοστώσει είναι ο μοναδικό τρόπο για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και στα διοικητικά συμβούλια. Συμφωνώ ότι τα πολιτικά κόμματα είναι το κλειδί για την επίλυση των προβλημάτων των γυναικών. Δυστυχώ δεν έχουμε ε, αρκετή δημοκρατία και στα πολιτικά κόμματα τα ίδια. Το δημοκρατικό λοιπόν έλλειμμα αυτό είναι πρόβλημα όχι μόνο στη Μολδαβία, αλλά και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Και θα ήθελα να σα ενθαρρύνω, πρέπει να επιδείξετε μεγάλο θάρρο και μεγάλη τόλμη για να περάσουν τα μέτρα αυτά. Θα πρέπει να έχετε αυτοπεποίθηση, θα πρέπει να αγωνιστούμε για τι ποσοστώσει, γιατί μου φαίνεται ότι είναι τρόπο τρόπος τελικά. Όταν μιλάμε για διαφασικούς μισθού για την ίση εργασία, θα πρέπει να το καταδικάσουμε αυτό. Δεν είναι δυνατόν οι γυναίκε και οι άντρε να μην έχουν την ίδια αμοιβή. Εγώ είμαι από την Κροατία. Στην Κροατία διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές ανισότητες, πολλές αδικίες. Και αυτό θέλουμε να το καταπολεμήσουμε μέσω του έργου μας στην Επιτροπή αυτή. Οι γυναίκες τώρα στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Είναι μεγάλο το επιδευμα αυτό της Επιτροπής μας, αλλά και της κυρίας Vivian Redding, η οποία κατάφερε να περάσει το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτό από το 30% για να πετύχουμε το 50%. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε. Συνδυασμό επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Πώ βρίσκει κανεί ε, την ισορροπία. Δεν είναι απλό. Και πολλά ε, εξαρτώνται από τι υποδομέ, την εξέλιξη των υποδομών στην ε, χώρα σα. Είναι θέμα, για παράδειγμα, παιδικών σταθμών, σχολείων, ε, φύλαξης. Και στο σημείο αυτό μεγάλο ρόλο παίζει και το ΑΕΠ της ε, κάθε χώρας, της οικονομική εξέλιξη, οικονομική πρόοδος της κάθε χώρας. Ε, θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε μια ίση δημοκρατική κοινωνία και στη Μονταβία και στην Κροατία και σε όλες τις χώρες θέλουμε να πετύχουμε την ισότητα τελικά. Βλέπουμε τι γίνεται και με τις γυναίκες μετανάστες και τις γυναίκες πρόσφυγες. Και είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ κάποια από τα καταλήμματα αυτά στη Μαβαρία, για παράδειγμα, στη Γερμανία, όπου και μετέβησα. Είδα ότι είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικές οι καταστάσεις και πραγματικά είναι πολύ καλός ο τρόπος διαβίωσης. Δεν είναι απλό όμως και από εμά εξαρτάται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να εκπροσωπούμε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι γυναίκες των γειτονικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προωθήσουμε την ισότητα. Δεν μιλάμε για απλό φεμινισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπήρχε από τις απαρχές του κόσμου. Η γυναίκα και ο άντρας σε ίσες θέσεις. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας λοιπόν σήμερα. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω κάποια μέλη της ε, Μολδαβικής Αντιπροσωπείας να πάρουν το λόγο για να απαντήσουν αν θέλουν. Είτε η Λιλιάνα ή κάποιος άλλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια εκτίμησης που ακούσαμε. Δεν μπορέσαμε σε μία μικρή εισαγωγή και παρουσίαση να καλύψουμε όλα τα ζητήματα αυτά που αναφέρετε. Αν σα ενδιαφέρει, ευχαρίστω να κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση. Εμεί είμαστε στη διάθεσή σας. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω και να κάνω κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά αυτά που είπε η κυρία Κοσλόφσκα. Ότι είναι καλύτερα να ακολουθήσουμε το μοντέλο τη Σουηδία, για να υπάρχει μια κανονική εκπροσώπηση χωρίς ποσοστώσεις και υποχρεωτικές ε, υποχρεωτικού όρου. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, η Σουηδία τα πέτυχε αυτά μετά από μια μεγάλη περίοδο διαρκούς αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτή την υψηλή εκπροσώπηση των γυναικών στο Κοινοβούλιο την πέτυχαν μετά από μια μακρά περίοδο αγώνα. Εμεί δεν έχουμε 50 χρόνια να περιμένουμε Θέλουμε τώρα να αλλάξει η κατάσταση και ο μοναδικό τρόπο να αλλάξει αυτό στο σύντομο χρονικό διάστημα είναι να εισαχθούν υποχρεωτικέ ποσοστώσει για τα πολιτικά κόμματα, για την υποχρεωτική εκπροσώπηση ανδρών, γυναικών και ανδρών, αν χρειαστεί. Αν υπάρχει δηλαδή υπερβολική εκπροσώπηση γυναικών σε κάποιο κόμμα, να σκεφτούμε και την ποσόστοση για του άνδρε. Ε, δεν φαντάζομαι αυτό να συμβεί στο εγγύη μέλλον στη Μολδαβία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό το θέμα το των στον ενδεχομένως να εισαχθεί ω μέτρο για 10-15 χρόνια μέχρι ότου αλλάξει η συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων και ενδεχομένως σε 15 χρόνια να αποφασίσουμε ότι δεν χρειάζεται πλέον το στοιχείο αυτό στην νομοθεσία μας. Αλλά έχουμε την κυρία Μπουλίγκα, την πρώην Υπουργό ε, Κοινωνική Προστασία. Έχει τεράστια εμπειρογνωμοσύνη και η κυρία Τσουμπέσκα έχει... είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, κοινωνικής προστασίας. Θα τι καλέσω λοιπόν να πάρουν το λόγο για να μας μιλήσουν για τις μισθολογικέ διαφορές, για τις διαφορές στην, ε, στον ύψο των συντάξεων. Μπουλίκα, κύριε Μπουλίκα λοιπόν και κύριε Ντομέκα για να μας ε, σχολιάσουν τα ζητήματα αυτά. Bună ziua! Stimată doamnă președinte, stimate colege... Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ ε, από πλευράς και των συναδέλφων μας για αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε μια συζήτηση στα πλαίσια της συνεδρίασης της Επιτροπής σας. Είδαμε πώς συζητάτε διάφορα θέματα ως Επιτροπή, θέματα που και εμάς μας απασχολούν ιδιαίτερα και είναι πολύ σημαντικά και αγαπητά και για μας. Ε, και η Ομολδαβία όπως ε, και άλλες χώρες της Ένωσης έχουν επικυρώσει πολλές συμβάσεις για θέματα γυναικών και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ειλικρινά και ανοιχτά αυτή τη συζήτηση. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε μόνο στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και για τη συμμετοχή του ε, στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών ζωής και, του, και εκδημοκρατισμού της χώρας τους. Όλα αυτά μας κάνουν να πιστεύουμε πολύ περισσότερο στον αγώνα μα. Στην Μολδαβία τα πολιτικά κόμματα και λόγω της δημογραφικής κατάσταση, γιατί 52% του πληθυσμού είναι γυναίκες και οι γυναίκες είναι πολύ ενεργές και κατά τις προεκλογικέ διαδικασίε και εκστρατείε. τα περισσότερα λοιπόν πολιτικά κόμματα στα προγράμματά τους και στους κανόνες διοντολογίας τους έχουν ποσοστώσεις για εκπροσώπηση των δύο φύλων και στα κόμματα και στις ε, δομές των κομμάτων, τα διάφορα όργανα. Όμως οι ποσοστώσεις αυτές ε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν έχουν δώσει και τόσο αξιόλογα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Οι γυναίκες ε, απλώς ήταν διακοσμητικές. Υπήρχαν δηλαδή κάποιες γυναίκες σε κάποια όργανα και σε, μεταξύ κάποιων εκλεγμένων εκπροσώπων. Αλλά ορισμένε μη κυβερνητικέ οργανώσει μα είπαν ότι πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικέ ποσοστώσει για τη συμμετοχή του και ε, σε πολιτικά όργανα και ε, στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Στο Κοινοβούλιο ε, της χώρας μας προωθούμε τρία νομοθετήματα που ασχολούνται με την καθιέρωση ποσοστώσεων και οι ποσοστώσεις αυτές είναι της τάξης του 30, 40 ή και 50%. Και στην πλατφόρμα μας ε, κάνουμε προσπάθεια για να προωθήσουμε ε, μια μεγάλη προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινή γνώμης και των πολιτικών κομμάτων για να στηριχθεί η τελευταία πρόταση νομοθεσίας που κάνουμε γι' αυτό. Στηρίζουμε λοιπόν όλες τις προσπάθειες τις οποίες και εσείς αναφερθήκατε. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να υπάρξει και η αναγκαία υποδομή για να βοηθήσουμε τις γυναίκες και για να αλλάξουν και οι για να μπορούν να συνδυάσουν καλύτερα οι γυναίκες την ε, οικογενειακή ζωή με την εργασία. Αλλά η έλλειψη των υποδομών είναι ιδιαίτερα ε, μεγάλος φραγμός για να μπορέσουν να συμμετάσχουν ε, οι γυναίκες είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε εθνικό επίπεδο στην πολιτική. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε πολλές πρωτοβουλίες για να καταργηθεί και αυτή η διαφορά στο επίπεδο αποδοχών. Γιατί έχουν υπάρξει και μελέτες που δείχνουν ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε επαρκής νομοθετική προσπάθεια για να επιβάλλει ίση αμοιβή για ίση εργασία για τα δύο φύλλα. Επίσης, ε, υπάρχει και διαφορά στην ηλικία συνταξιοδότηση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πέντε ε, χρόνια είναι αυτό, αυτή η διαφορά της ηλικίας Τα Θεωρούμε ότι αυτό είναι τεράστια ε, ε, ανισότητα μεταξύ των φίλων. Προσπαθούμε να αλλάξουμε την ομοθεσία για παράδειγμα για την γονική άδεια να μπορούν να λάβουν και οι, γονείς, και, συγγνώμη, και οι πατέρες γονική άδεια. να μπορούν όπως έλεγα και οι πατέρες να έχουν 14 μέρες γονική άδεια, πατρική άδεια λοιπόν. Αμέσως μετά τον τοκετό, τη γέννηση του παιδιού. Γιατί μπορούν να λάβουν ε, γονική άδεια για την ε, ανατροφή μετά των παιδιών. Ήδη οι πατέρες και μπορούμε να σας ε, διαβεβαιώσουμε ότι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αλλάζει σιγά σιγά η αντιμετώπιση και η νοοτροπία. Είναι σημαντικό λοιπόν να ακούσουμε και ποια είναι τα προβλήματα που εσείς αντιμετωπίσατε, πώς τα αντιμετωπίσατε, γιατί η πείρα σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί έτσι θα βελτιωθεί και η δυνατότητα λειτουργίας και αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας αυτής που έχουμε δημιουργήσει, γιατί θεωρούμε ότι ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο ανήκουμε, θα πρέπει να ακούγεται ξεχωριστά η φωνή μας. Πρέπει ε, όχι απλώς να παρακολουθούμε, αλλά να συμμετέχουμε. Θέλουμε επίσης ε, στη Μολδαβία να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να γίνει εθνική νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία, για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των γυναικών, είτε στις αστικές περιοχές, είτε στην Ήπεθρο, όπου και αν εργάζονται, είτε εργάζονται ως υπάλληλοι, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες, αυτή είναι η κοινή στόχη ε, γύρω από τους οποίους ε, έχουμε συσπηρωθεί και εργαζόμεθα ενωμένε και το γεγονός ότι μπορούμε να σας μιλήσουμε για το θέμα αυτό μας βοηθάει να αποκτήσουμε και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Η κυρία Ντομέντη θα πάρει τώρα το λόγο που είναι επικεφαλής της Επιτροπής για Κοινωνικές Υποθέσεις ε, στο Κοινοβουλίο μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε για συμμετοχή στη συνεδρίαση αυτή. Τα ζητήματα που θίξατε και η προσέγγιση είναι τα ίδια. Εδώ στη χώρα μας ίσως να είναι πιο σοβαρά, τα, σοβαρή η κατάσταση από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όμως δεν πάβουν να είναι τα ίδια ζητήματα που μας απασχολούν. Εάν ε, σκεφτούμε την ε, διακρίσεις κατά των γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες, οι διακρίσεις υπάρχουν όσον αφορά τη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, υπάρχει και εδώ στη διαφορά μάλλον μισθών, αλλά και ασφάλισης. Υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορές και ακόμα και αν η νομοθεσία δεν περιλαμβάνει ρητά αυτές τις διακρίσεις, υπάρχουν στην πράξη. Στατιστικώς η γυναική μισθή είναι γύρω στο 20% ε, χαμηλότερη από τον ανδρών. Και αυτό εξηγείται καταρχά από το γεγονός ότι οι γυναίκες εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς από τους άντρες και αυτό είναι το ίδιο πρόβλημα παντού. Οι γυναίκες επιλέγουν δικαιοκότητες και επαγγέλματα τα οποία δυστυχώς δεν αμείβονται τόσο καλά όσο αυτά των αντρών. Είτε είναι στην εκπαίδευση, είτε είναι η κοινωνική πρόνοια, η κοινωνική λειτουργία κτλ. Και στην ε, Μολδάβα οι κοινωνικές ε, δομές δεν είναι τόσο καλά ε, οργανωμένες, οπότε οι γυναίκες φέρουν το βάρος της φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ανθρώπων με αναπηρίες στην οικογένεια και αυτές οι δραστηριότητες είτε αμείβονται πολύ πενιχρά ή και καθόλου γιατί πολλέ φορέ δεν υπάρχουν προβλέψεις και οι γυναίκε οφείλουν να κάνουν αυτές τις ε, ε, δραστηριότητε, Δεν μπορούν να, δηλαδή να φροντίζουν ηλικιωμένα σε παιδιά, δεν μπορούν να εργαστούν αλλιώς ή λείπουν από την αγορά εργασία για πολύ καιρό και μετά πολύ δύσκολα μπορούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασία. Προσπαθούμε λοιπόν μέσω διαφόρων προγραμμάτων να βοηθήσουμε τις γυναίκες ώστε να επανέλθουν στην αγορά εργασίας αφού έχουν φροντίσει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Επίσης προσπαθούμε να προσανατολίσουμε τις γυναίκες σε τομείς όπου παραδοσιακά είναι ε, ανδρικά επαγγέλματα όπως η αρχιτεκτονική ή η πολεοδομία. Μιλούσατε για τις συντάξεις και την κοινωνική ασφάλιση και εμείς εδώ έχουμε ένα κενό το οποίο εξαρτάται και από τους μισθούς εφόσον η μισθή είναι χαμηλότερη και τελικά η σύνταξη είναι πολύ χαμηλότερη. Έχουμε και ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες και αυτό είναι το πρόβλημα των μεταναστών, των όσων έφυγαν από τη Μολδάβα για να εργαστούν αλλού, στη Δύση και στην Ανατολή όπου πολλοί επανέρχονται στην Μολδάβα, ωστόσο δεν έχουν αρκετά χρόνια εργασίας ώστε να μπορούν να λάβουν πλήρες συντάξει. Και αυτή τη στιγμή η Δημοκρατία της Μολδάβα δεν έχει συνάψει συμφωνίες περί κοινωνικής ασφάλισης είναι πολλές χώρες, οπότε πολλές χώρες μπλοκάρουν ή αρνούνται το διάλογο με τη χώρα μας, δεν θέλουν να υπογράψουν αυτές τις συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και άλλα φόρα καθώς χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία συνυπογραφής κοινωνικών συμφωνιών ώστε τα κοινωνικά δικαιώματα εργαζομένων της Μολδάβας σε άλλες χώρες να αναγνωρίζονται και όταν, ακόμα και όταν αυτοί επιστρέφουν στην ε, χώρα τους. Τώρα, για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια δεν έχουμε διακρίσει σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν γυναίκες, πολλές μορφωμένες γυναίκες που έχουν ε, διοικητικές ε, θέσεις και μάλιστα εκτιμώνται πολύ στην καθημερινή τους εργασία, αλλά βεβαίως για να γίνει αυτό έχουμε εισάγει αλλαγές και στην ίδια την νομοθεσία μας. όσον αφορά την άδεια πατρότητας. Και οι δύο γονείς και οι παππούδες έχουν τη δυνατότητα με βάση την νομοθεσία να φροντίσουν τα παιδιά. Και αυτό το χρησιμοποιούν πολλοί οι γυναίκες, ε, αυτό το στο δικαίωμα. Τέλος, θέλω να πω ότι όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αν χρησιμοποιούμε μόνο τις ποσοστώσεις ως απέτηση, δεν πρόκειται αυτό να αποτελέσει επαρκή λύση. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσεται και μια θετική εικόνα των γυναικών στην πολιτική της εργασίας μας, δηλαδή στο Κοινοβούλιο και προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε, πολύ, είμαστε πολύ δραστήριες. Οι γυναίκες βουλευτές έχουν το μεγαλύτερο ρυθμό πρωτοβουλειών και πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες έχουν ήδη εγκριθεί. Μέσω αυτών δε θέλουμε να στηρίξουμε την περαιτέρω συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η εκπρόσωπο ε, τη ε, Μολδαβική ε, Βουλή. Αν έχετε άλλε ερωτήσει, ευχαριστώ να τι απαντήσουμε, αλλά δεν θέλω να μονοπολίσουμε. Σα ευχαριστώ, η Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πραγματικά. Ευχαριστώ όλους τις εκπροσώπους του Μολδαβικού Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι από τη Λιθουανία. Κατανοώ λοιπόν πολύ καλά την τοποθέτησή σας και τη θέση σας. Εύχομαι ειλικρινά να επικρατήσει η διαδικασία εκδημοκρατισμού στη Μολδαβία και η ισότητα των φίλων να καταστεί κάτι αυτονόητο. Ένας στόχος ε, αυτονόητος. Πρωτού εκλεγώ βουλευτής, ήμουν υπουργό εργασία και Κοινωνικής Ασφάλειας στην ε, Λιθουανία. Θυμάμαι πολύ καλά λοιπόν όταν συζητούσαμε την, ε, το ενδεχόμενο νομικής κατοχήρωσης της ε, γονικής άδεια, Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι συζήτηση χρειάστηκε, τι διαπραγμάτευση χρειάστηκε και τώρα μετά από λίγα χρόνια αυτό θεωρείται κάτι εντελώς φυσιολογικό, κάτι αυτονόητο, αποδεκτό. Και πολλοί άνδρες χρησιμοποιούν αυτά, αυτή τη γονική άδεια. Εκπρόσωπο λοιπόν τους σοσιαλιστές στην ε, χώρα μου και έχουμε ποσοστώσεις λοιπόν για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Ανάλογα με το που γίνονται οι εκλογές, αν είναι για στο δημοτικό επίπεδο ή στο βουλευτικό επίπεδο. 40 έως 60%. Και τηρείται λοιπόν αυτή η ποσόστοση. Και το εκλογικό κοινό όμως υποστηρίζει το σύστημα αυτό. Έχουμε 11 μέλη από την Λιθουανία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ είμαι η μοναδική γυναίκα. Πραγματικά στο αυτό. Παρά το γεγονός μάλιστα ότι στους κατάλογους, καταλόγους υποψηφίων συμπεριλήφθησαν πολλές γυναίκες. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει η κατάσταση και στους ε, διάφορους ε, τομείς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εργασία με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Σε όλους αυτούς τους τομείς θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε για τη λήψη αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα το συνδυασμό επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και πάλι την αντιπροσωπεία σας από πλευρά τη Επιτροπή μα. Σας εύχομαι κουράγιο, υπομονή και επιμονή, γιατί τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν. 25 χρόνια, ξέρετε, δεν είναι μεγάλη περίοδος στην εξέλιξη ενός κράτους, ενός εθνούς και η αλλαγή νοτροπίας απαιτεί χρόνο. Φυσικά η παιδεία αποτελεί ζήτημα κλειδί και μάλιστα από τις νεαρότατες ηλικίες. Θα πρέπει τα παιδιά να γνωρίζουν, να τους εξηγείτε τι είναι η ισότητα των φίλων και τι μπορεί να έχει ως συνέπεια για το κράτος και για τον λαό. Θεωρώ ότι θα είναι υποφελής η ανταλλαγή αυτή απόψεων. Θα μας ωφελήσει και εμάς, στην Επιτροπή μας, όταν θα καταρτήσουμε γνωμοδότηση για την κατάσταση των γυναικών σε χώρες Ανατολικής Γειτονίας. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στο έργο σας. Ναι, κοιτάξτε, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλες τις αντιπροσωπείες μας, να σας προτείνω αν ε, χρειάζεστε πιο πολλές πληροφορίες για τα ζητήματα επί των οποίων εργάζεται η Επιτροπή σας, είμαστε πρόθυμες ασφαλώς να σας παρέχουμε τις ειδικές πληροφορίες. Ε, στείλτε μας τις ερωτήσεις ε, για τις οποίες θέλετε στοιχεία και ευχαρίστω θα τις απαντήσουμε. Σας ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι η συγχύτρια σίγουρα θα λάβει υπόψη την γενική αυτή πρότασή σας και μια και έτσι ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη και δεν έχουμε άλλα στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, όσοι συμμετείχαν. Ε, γενικά η πρόεδρος ευχαριστεί και την Τερμινής. Και ζητώ συγγνώμη που ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση και μία ώρα νωρίτερα. 22 και 23 Μαρτίου η επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.